Eh, Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την ε, προσέλευσή σας και την συνέπεια. Έχουμε κάποια κενά στα έδρανα, όμως δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε την ελβετική συνέπεια της Προέδρου της Ελβετικής Νομοσπονδίας, Μισλίν Καλμιρέη, η οποία ήταν στην ώρα της και δεν θέλουμε να την καθυστερήσουμε περιμένοντας εμείς να ξεκινήσουμε. Μαζί μας είναι και η νεότατη πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ελβετικού Εθνικού Συμβουλίου, κυρία Μάρκ Μπάλτερε και άλλα μέλη της Ελβετικής Αντιπροσωπείας. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας συναντώ, κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία ανέκαθεν είχαν στενούς δεσμούς, ανέκαθεν συμμερίζονταν τις ίδιες αξίες και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία μπορούν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν κοινέ προκλήσεις. Βεβαιότατα η επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συνοδεία κάποιων προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπους από τη δική μας επιτροπή, ο κύριος Προβέρα, ο πρώτος αντιπρόεδρος. Όλα αυτά πιστοποιούν το μεγάλο ενδιαφέρον μας και τους κοινούς μας στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται κάποιες στατικές προτεραιότητες με την Ελβετική Συνομοσπονδία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τον Νότιο Κάφκασο, το Ιράν, το Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική ως γεωγραφικές περιοχές. Ιδίως ό,τι φορά τη Βόρεια Αφρική γνωρίζω ότι με την ε, Υπουργηγό Εξωτερικών μας, την κυρία Άστον, βρίσκεται στην Τίνιδα τον περασμένο μήνα στα πλαίσια της ομάδας δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την Ισία Και ο συνάδελφος Αλαφράγκα, ο κ. Παντσέρη, ο πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας για το Μακρέβο, ο κ. Νέιτ, που εκπροσωπεί την ομάδα των φιλελευθέρων, συμμετείχαν στην επίσκεψη. Η χώρα σας λοιπόν στηρίζει την δημοκρατική μετάβαση των Αράβων γειτόνων μας, και αυτό βεβαίω είναι κάτι που όλοι το εκτιμούμε ιδιαίτερο γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν θέλω να σας κλέψω άλλο χρόνο από την ομιλία σας. Θα συζητήσετε και με του συναδέλφου σα ευχαριστώ ξανά για την προσέλευσή σας και θα σας ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ ίδιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας ε, με τιμά. Με προσκαλέσατε να μιλήσω ενώπιον της τόσο σημαντικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ελβετίας. Η Ελβετία από πολλές πλευρές είναι στενά συνδεδεμένη με πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής όσο και τα λοιπά ε, κράτη-μέλη μεταξύ τους. Επί σειρά ετών αναπτύξαμε διάφορες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 120 διμερείς συμφωνίες υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία, εκ των οποίων 20 πολύ σημαντικές. Η Συμφωνία Σέγγεν, Συμφωνία για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Προσώπων και Αυτές οι σου σχέσεις ε, δεν μπορούν ε, να συγκριθούν με άλλες σχέσεις που έχουμε με τρίτες χώρες σε καμία περίπτωση. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι τρίτη χώρα η Ελβετία και ανήκει στο ε, φάσμα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την οποία εξωτερική πολιτική έχει ευθύνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πρέπει να εγκρίνει και να επικυρώσει τις συμφωνίες που συνάπτονται με την Ελβετική Ομοσπονδία. Ε, εξού και η παρουσία μου εδώ. Θα ήθελα να κάνω δύο προκατακτικές παρατηρήσεις. Ε, πρώτον, για τις σχέσεις της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρετε και δεν χρειάζεται να επιμείνω σε αυτό το θέμα. Κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τις παγκόσμιες σχέσεις δυνάμεων. Ε, σήμερα οι βιομηχανοποιημένες χώρες ε, έχουν ένα μερίδιο στην παγκόσμια ανάπτυξη από το 1980 μέχρι τις αρχές του 2000 από το 60 με το 30% και την ίδια περίοδο τριπλασιάστηκε σχεδόν το ποσοστό στην παγκόσμια ανάπτυξη που αντιστοιχεί στην Ασία. Αυτό καταδεικνύει ότι η προεξάρχουσα θέση που είχε η Δύση στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων ε, που ήταν, ε, είχε πάγιο χαρακτήρα υπό διαφορετικές μορφές ήδη από τον 18ο αιώνα φτάνει στο ε, τέλος της. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση, σήμερα ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κείμενο με παγκόσμιου ε, κινδύνους, ε, παγκοσμιοποιημένους κινδύνους, η τρομοκρατία, φερρυπίν, ε, κλιματικές αλλαγές, μεταναστευτικές ροές. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να βρουν απάντηση από τη δράση ενός μόνο κράτου, ακόμη και είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη. Άρα σε πολυμερές επίπεδο θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις εργασίες μας και η μολυμερής διάσταση της διακυβέρνησης ε, είναι η μόνη που θα φέρει απαντήσεις ε, στα πλαίσια εταιρικών σχέσεων με άλλα κράτη-μέλη. Η απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρος σε αυτές τις προκλήσεις είναι η ολοκλήρωση, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση η Ενωμένη Ευρώπη θεωρεί ότι είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί ε, σε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελβετία είναι μόνη, δηλαδή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα στη σημερινή μου ομιλία να σας ε, εξηγήσω πώς αντιμετωπίζουμε εμείς αυτή την νέα κατάσταση, τα νέα δεδομένα, με ποιο τρόπο προσπαθούμε να ε, αυξήσουμε την επιρροή που έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, δηλαδή την ασφάλεια και την ευημερία των Ελβετών πολιτών. Πρώτος άξονας ε, της πολιτικής μας είναι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δεύτερος άξονας της πολιτικής ε, είναι η ε, διερεύνηση ε, ενδυνάμει προνομιακών εταιρικών σχέσεων, στρέφοντας το βλέμμα μας κυρίως προς την Ανατολή και δεύτερος άξονας η θέση της Ελβετίας στα πλαίσια της πολιτικής, της ειρηνευτικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής. Ας αρχίσουμε με τον πρώτο άξονα, δηλαδή σχέσεις Ελβετίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελβετία ακολουθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική, ούσα μέλος ε, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, του ΟΣΑ, της ΕΖΕΣ συμμετέχουμε στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας αυτόνομης συνεισφορά προ τα κράτη-μέλη που προσχώρησα μετά το 2004 επενδύουμε πάρα πολύ σημαντικά κονδύλια άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για την οικοδόμηση ε, των εγκαρσίων σιδηροδρομικών συνδέσεων μέσα από τι Άλπεις για να διευκολυνθεί μεταφορά των εμπορευμάτων από το βορρά προς τον νότο τη Ευρώπη και ε, ε, συμμετέχουμε επίσης στην ευρωπαϊκή πολιτική, στην Βαλκανική Χερσόνησο. Είμαστε παρόντες με όλα τα μέσα που έχουμε ε, για την αμυντική μας πολιτική και την εξωτερική μας πολιτική στο Κωσυφοπέδιο και το είπατε και εσείς Πρόεδρε στην Βόρειο Αφρική όπου ήδη από τα πρώτα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης ε, προσέφερε η Ελβετία ανθρωπιστική βοήθεια και σήμερα δίνει βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης ε, σε αυτές τις χώρες, ε, κυρίως ενθαρρύνοντας ε, την ίδρυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη δράση τους, ε, καθώς ε, και την, σχετικά με την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην ηγεμόνων αυτών των χωρών. Επίσης, η Ελβετία σε αυτό το τομέα έχει ρόλο πρωτεργάτη. Θα ήθελα να το τονίσω. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπα και προηγουμένως, έχουμε 120 διμερείς συμφωνίες και αυτό το σύστημα sui generis που αναπτύχθηκε επί διμερούς βάσεως ε, ε, υπακούει φυσικά στις επιταγές του ε, διμερισμού, ας το πούμε στις διμερούς διάστασης. Δηλαδή, συνήψαμε συμφωνίες σε διάφορους τομείς, όμως στην τράπεζα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τίθενται τώρα κάποια θεσμικά ζητήματα. Θέλουμε να εισέλθουμε σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων ε, για κάποιες ε, πολύ ουσιαστικέ συμφωνίες, παραδείγματο χάρη για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τις ελεύθερες ε, συναλλαγές στη Γεωργία, στη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα Γαλιλαίο, διάφορα κοινά προγράμματα που θα θέλαμε να φέρουμε σε πέρας. Για τα θεσμικά ζητήματα να προσθέσω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι στους τομείς όπου η Ελβετία έχει πρόσβαση στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της και τις μελλοντικέ αλλαγές ε, του ενωσιακού δικαίου, του δικαίου της Ένωσης. Φυσικά προτιθέμεθα να το κάνουμε υπό την αίρεση του σεβασμού της κυριαρχίας ε, της Ομοσπονδίας μας. Δεν θέλουμε αυτά να γίνονται με αυτόματο τρόπο, αλλά να ακολουθούνται οι ελβετικές νομοθετικές διατάξεις. Πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα ζητήματα, ε, όπως παραδείγματος χάρη εφαρμογή των συμφωνιών ε, Ελβετίας-Ευρωπαϊκής Ένωση όταν ε, σχετίζονται με την, τα θέματα ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας παραδείγματος χάρη ή της επίλυσης των διαφορών. Κάνουμε διερευνητικές συνομιλίες προς το παρόν. Ε, πάντως η Ελβετία το ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστροφο φυσικά ισχύει. Η Ελβετία, ε, ο οικονομικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δεύτερος οικονομικός εταίρος της Ένωσης μετά τη ΣΥΠΑ, είναι επίσης ε, ο δεύτερος πελάτης της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποδέκτης ε, του 60% των εξαγωγών μας και 80% ε, των εισαγωγών μας με ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο ε, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ύψους 24 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων περίπου. Για την εξωτερική πολιτική ε, υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους τομείς, συμβαδίζουμε, συνεργαζόμαστε και θα αναφερθώ σε αυτούς μεταγενέστερα. Για το δεύτερο σημείο, Ε, όταν σας έλεγα ότι στρέφουμε το βλέμμα μας προς ε, Ανατολάς, η Ελβετία ε, πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι άλλαξαν άλλαξε η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων και θα πρέπει να τροποποιήσουμε και να αυξήσουμε την εκπροσώπησή μας στην Ανατολή. Ανοίξαμε διάφορα προξενία και ε, ε, διπλωματικές αποστολές και από το 2005 επιθυμούμε να έχουμε ε, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με διάφορους παγκόσμιους παίκτες, είπα παραδείγματος χάρη Ρωσία, ε, Νότιος Αφρική, Βραζιλία και σίγουρα παραβλέπω και κάποιους. Ε, ε, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. και ενισχύουμε αυτές τις στρατηγικές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου. Το όραμα αυτό μας επιτρέπει να προωθήσουμε φυσικά και τις εξαγωγές μας σε αυτές τις χώρες. Κατόπιν για το τρίτο σημείο ε, που σχετίζεται με τη θέση της Ελβετίας ως προς τις ειρηνευτικές διαδικασίες και την αναπτυξιακή πολιτική σε διεθνή κλίμακα, ε, θελήσαμε ε, να αναδείξουμε την Ελβετία σε παγκόσμια φορέα που χαρακτηρίζεται από την περιβόητη ουδετερότητά μας. Ε, στην παγκόσμια σκηνή ε, θεωρείται ότι η Ελβετία δεν έχει κρυφό πρόγραμμα, ε, ε κρυφό δηματολόγιο. Ε, επίσης θεωρείται ότι είμαστε αντικείμενοι και ε, ε, θέλουμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες ε, του διεθνούς δικαίου στα ανθρωπιστικά ζητήματα όσο και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Προσωπούμε τα φέροντα της Γεωργίας στη Ρωσία ε, και κάναμε μια διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Αρμενία και την Τουρκία για την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων αυτών των χωρών που υπέγραψαν τα πρωτόκολλα της Ζηρίχης ε, το 2009 και τώρα συνεχίζουμε την επιδιαιτησία που έχουμε αναλάβει με, ανάμεσα στη Γεωργία και τη Ρωσία ε, για την ε, ε, είσοδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου της Ρωσίας. Και άλλες επιδιαιτησίες συνεχίζονται. Θα ήθελα να αναφερθώ στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η Ελβετία στην Μέση Ανατολή. Η Ελβετία εκεί δεν έχει ρόλο στρατηγικού εταίρου. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφοροποιημένο ρόλο σε σχέση με το δικό μας, ε, διότι πρόκειται για ε, παγκόσμιο εταίρο, γιατί ανήκει στο κουαρτέτο, σε αυτή την τετραμερή δύναμη, ενώ η Ελβετία όχι. Στη Μέση Ανατολή λοιπόν δραστηριοποιούμαστε για να προαγάγουμε το διεθνές δίκαιο για τα ανθρωπιστικά ζητήματα, για να αποφευθούν οι παραβιάσεις ε, του διεθνούς δικαίου. Επίση ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός. Ε, από αυτή την πλευρά υποστηρίξαμε μια ιονή συμφωνία ανάμεσα ε, στην Ισραηλινή και την Παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για την πρωτοβουλία της Γενέβης. Ε, και δημοσιεύτηκαν τα τελευταία πρακτικά σε σχέση με την ασφάλεια στην περιοχή. Το καλοκαίρι που μας πέρασε είναι ένα έγγραφο που περιέχει σχεδόν το 90% των ε, λύσεων που ενδεχομένως θα συμπεριληφθούν σε ένα μελλοντικό ειρηνευτικό σχέδιο. Το πρόβλημα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ε, στη Μέση Ανατολή να προσέλθουν ναι, ε, οι εμπλεκόμενοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ιδού. Δεν θέλω στην παρουσίασή μου να μακρηγορήσω και με τα χαράς να απαντήσω και να επανέλθω σε διάφορα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν μετά από τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη ορισμένους συναδέλφους που έχουν ζητήσει να παρέμβουν και πρώτος θα είναι ο κύριος Σφόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε και εσάς κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση των κυριότερων στόχων σας. Ως Αυστριακός εξακολουθώ να εκφράζω την θλίψη μου που η Ελβετική Ομοσπονδία δεν εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα με ενδιαφέρουν προκειμένου τώρα δύο πράγματα. Πρώτο, που βλέπετε το μεγαλύτερο περιθώριο για βελτίωση και πιο στενή συνεργασία ακόμη μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τώρα της εντάξεως που θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν. Η δική μου εμπειρία από την ελβετική πολιτική είναι ότι έχει δραστηριοποιηθεί πολύ, ιδίω υπό την δική σας ε, ηγεσία, και συνεργάζεται πολύ πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ αν έχετε κάποιο όραμα για το ποιο μπορεί να είναι το δεύτερο βήμα μετά από αυτό. Ένα άλλο θέμα τώρα λιγότερο εύθυμο, το τραπεζικό απόρριτο της ε, ε, Ελβετίας. Και η δική μου χώρα είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που έχει ακόμη το τραπεζικό απόρριτο, εγώ βέβαια διαφωνώ. Έχετε μια συμφωνία με την Γερμανία που από όσο γνωρίζω ακόμα ε, δεν έχει προχωρήσει στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα θεωρούν ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι διότι καλούνται να πληρώσουν ακόμα περισσότερα Περισσότερου φόρου και κερδίζουν λιγότερα, ενώ οι πλούσιοι πήγαν τα λεφτά του απλώ στην Ελβετία. Έχει λοιπόν εν τέλει ως στόχο το τραπεζικό απόρριτο την προστασία των πλούσιων και των μηχανογραφιών τους. Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο και γι' αυτό η ερώτησή μου προς εσάς. Πώς το βλέπετε το θέμα αυτό, πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε, να αποκρούσετε το επιχείρημα πολλών Ελλήνων ή θεωρείτε κι εσείς ότι όντως έγκαιρα πολλοί Έλληνες μετέφεραν τα στοιχεία του ενεργητικού τους στην Ελβετία. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ. Ο κύριος Παντσέρη χρειάστηκε να βγει για λίγο. Αλλά είναι εδώ, τώρα μπορώ να του δώσω μέσα το λόγο. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, λέει ο κ. Παντσέρη. Εκείνο μίλησε εξ ονόματο των Δημοκρατών, εγώ θα μιλήσω εξ ονόματο των Σοσιαλιστών. Καλά λοιπόν, σα ευχαριστώ πρώτα για την έλευση σα εδώ, κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει, αν με επιτρέπετε. Άλλωστε, είναι και μεγάλη χαρά που σα βλέπω μετά από την Τίνιδα, δύο προ εβδομάδων την Τίνιδα είχατε φανεί πρόθυμοι να συνεργαστείτε για να γίνουν οι αλλαγές, να βοηθήσετε, να συμβάλλετε να γίνουν οι αλλαγές στην Βόρεια Αφρική, όχι μόνο σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και με την χορήγηση χρηματοδοτήσεως ή με την επιστροφή χρημάτων που υπό το δικτατορικό καθεστώς Μπεναλή είχαν εξαχθεί σε διάφορες χώρες και μεταξύ αυτών και στην δική σας. Δείξατε λοιπόν μια προθυμία να προωθήσετε αυτή τη διαδικασία, καθώς επίσης να προσφέρετε υποστήριξη και στην νομοθετική διαδικασία. Ποια θα είναι, τι, θα πράξετε εσείς νομοθετικά για να επιστρέψετε τα χρήματα αυτά στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Και δεύτερο, Γνωρίζετε ότι ένα από τα κέρια προβλήματα στις σχέσεις μας με τον Νότο είναι η κινητικότητα. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Η χώρα σας, εάν θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία της, που τόσο συχνά μιλάτε για αυτήν, θα ήταν διατηρημένη άραγε η Ελβετία να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθεί μια νέα διαδικασία ας πούμε, κινητικότητας η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χωρών του Νότου. Για την ώρα οι προσπάθειες αυτές δεν είναι ιδιαίτερα συντονισμένες. Φαίνεται δε πως αποτελούν ένα από τα θεμελιώδη θέματα για το μέλλον. Είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε λοιπόν θέματα κινητικότητας από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στην Πρόεδρο για να γίνει πιο ευθύς ο διάλογος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στον κύριο Σφόμποδα και στον κύριο Παντσέρη πρώτα για την Βόρεια Αφρική πιο γενικά και θα επανέλθω μετά για τα χρήματα των ηγετών τους. Για τα θέματα της Βόρειας Αφρικής. Οι εξεγέρσεις που έγιναν στην νότια ακτή Τη Μεσογείου έχουν βέβαια επιπτώσει και σε εμά, όπω έχουν και επιπτώσει στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπήρξε για μα πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε γρήγορα. Η σχέση τη Ελβετία δεν ήταν ιδιαίτερα ε, θετικέ με το καθεστώ Μπεναλί διότι είχαμε επικρίνει το καθεστώ αυτό για την έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών το 2005, ιδίω για την έλλειψη ε, ελευθερίας έκφρασης και ήταν βέβαια πάρα πολύ αρνητικές οι αντιδράσεις της τότε την Ισιακή εξουσίας. Με την, Λιβύα, με τη Λιβύη συγγνώμη, οι ε, σχέσεις μας ήταν ανύπαρκτες. Θα γνωρίζετε ίσως και τις περιπέτειες των Ελβετών ομήρων στην Λιβύη, ε, όπου τελικά οι σχέσεις μας και εμπορικές αλλά και ανθρώπινες είχαν φτάσει σχεδόν στο μηδέν. Και γι' αυτό αντιδράσαμε σχετικά γρήγορα στις ε, εξελίξεις που σημειώθηκαν σε Αίγυπτο, Λιβύη και την Ισία και αντιδράσαμε όχι μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και με τη βοήθεια όπως σωστά είπατε και στη δημιουργία ε, απασχόλησης επίσης ε, για την ρύθμιση των μεταβατικών θεμάτων και βεβαίως για την επιστροφή των χρημάτων των δικτατόρων. Γιατί? Γιατί η Ελβετία θεωρεί ότι τα χρήματα αυτά δεν τις ανήκουν. Έχουμε την θέληση να τα επιστρέψουμε το δυνατόν συντομότερο ε, στους ανθρώπους που τους ανήκουν. Άλλωστε δεν πρόκειται για νέα ε, στάση της ε, Ελβετίας. Έχουμε μάλιστα πρωτοποριακό ρόλο παίξει στην επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους. Έχουμε και από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Οι τράπεζες αλλά και οι διαμεσολαβητές όχι μόνο οφείλουν να γνωρίζουν το όνομα του ε, δικαιούχου του λογαριασμού, αλλά και αυτών που έχουν ε, οικονομικά το δικαίωμα στα χρήματα αυτά. Και αυτό είναι δύσκολο. Εφόσον υπάρχουν υποψίες, οι υποψίες αυτές πρέπει να ανακοινώνονται και λαμβάνονται μετά. Το δεύτερο θέμα είναι μπλοκάρισμα, κατάσχεση, επιστροφή των χρημάτων. Για τα καθεστώτα Μπέναλι, Μουμπάρακ, Καντάφη, εμείς μπλοκάραμε τα χρήματα αυτά ταχύτατα ώστε να μην μπορέσουν να μεταφερθούν σε άλλες ε, χώρες. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν μπλοκαριστεί. Δεν σημαίνει ακόμα ότι έχουν κατασχεθεί τα χρήματα αυτά. Η κατάσχεση πρέπει να περάσει βέβαια πρώτα από τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες. Είμαστε κράτος δικαίου. Αυτές οι διαδικασίες βέβαια ενδέχεται να απαιτήσουν χρόνο πλοίωνα των ορισμένων μηνών. Και γι' αυτό στον τομέα αυτό για τα θέματα μάλλον του τομέα αυτού. Πήγα και στην ε, Τίνιδα, μέσα στα πλαίσια της ε, Task Force Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ελβετίας, για να εξετάσουμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά τα οποία είχαν μπλοκαριστεί σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και σε άλλες χώρες, να επιστρέψουν το δυνατόν συντομότερο. Πρόσφατα εγκρίναμε ένα νόμο στην Ελβετία για να επιστραφούν χρήματα όταν δεν, υπήρχε, σαφή, δεν υπήρχαν σαφείς αποδείξεις για, τον προορισμό, για την ε, ε, πηγή τους. Ζήτησε και η Τινησία αυτό από την Ελβετία. Εμείς συνεργαστήκαμε με την Τινησία ώστε τα αιτήματα αυτά να ικανοποιηθούν και η συνεργασία αυτή να επιταχύνει τα πράγματα. Βέβαια, παραμένουν μακρόχρονες οι διαδικασίες και ένας από τους τρόπους που έχουμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες θα είναι να περάσουμε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα προχωρήσει σε κατάσχεση των χρημάτων αυτών και θα μας επιτρέψει έτσι να τα επιστρέψουμε. Αυτό έγινε στην περίπτωση της Λιβύης για τα ε, χρήματα ορισμένων κρατικών ε, φορέων ε, λιβικών. Υπάρχει τώρα και η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών που ε, επιλαμβάνεται του τους. Τώρα για την Αίγυπτο και την, ε, την Ισία όχι. ένα τρόπος εκεί για να επιταχυνθούν τα πράγματα θα πρέπει να είναι ίσως ο ίδιος δρόμο όπως έγινε δηλαδή για την Λιβύη δηλαδή να περάσουμε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που θα επέτρεπε κατάσχεση και επομένω μετά επιστροφή των χρημάτων. Η Ελβετία δεν έχει κανένα ιδιαίτερο συμφέρον να διατηρηθούν τα χρήματα αυτά στις τράπεζές της. Και γι' αυτό παίξαμε και ρόλο πρωτοπόρου από τα 5 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα τα οποία επεστράφησαν στις ε, ε, χώρες από τις οποίες είχαν προέλθει, η Ελβετία έχει επιστρέψει 1,7 δις. Και το μεγαλύτερο, 800 εκατομμύρια, στο Ταμείο Αμπασά στην Νιγηρία. Αυτά σχετικά με τα χρήματα των διαφόρων καθεστώτων, καθώς και για την παρέμβασή μας στην Βόρεια Αφρική. Ο κ. Φόμποντα με ρώτησε επίσης σε ποιον τομέα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε καλύτερα στην εξωτερική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απήντησα ήδη για τα θέματα της Βόρειας Αφρικής. Θα απαντήσω και για τα Βαλκάνια. Εδώ υπάρχει συνεργασία στην EULEX συμμετέχουν Ελβετοί ειδικοί στην EULEX στο Κόσοβο. Έχουμε και μια σημαντική κοινότητα στο έδαφος μας που προέρχεται από την πρώην Ιουγκοσλαβία, κάτι το οποίο εξηγεί βέβαια και το ενδιαφέρον της Ελβετίας για την ε, περιοχή αυτή της Ευρώπης και εξηγεί επίσης και ε, τον λόγο των δραστηριοτήτων μας και της στενής συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, χώρες αυτές. Η Ελβετία έχει λοιπόν πολιτική γειτονία και με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής αλλά και με την Ουκρανία καθώς και με άλλες χώρες που βρίσκονται ε, όμορες με τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν συγκλίνοντα συμφέροντα και εργαζόμαστε πραγματικά πολύ στενά. Συνεργαζόμαστε μάλλον το άλλο θέμα, για το τραπεζικό απόρριτο, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον να διατηρούμε στην Ελβετία χρήματα, κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από ροφοδιαφυγή στις χώρες τους. Και για τον λόγο αυτό εγκρίναμε, δεχθήκαμε τις προδιαγραφές του ΟΣΑ το 2009 σε ό,τι αφορά τις ε, σχετικές κοινοποιήσεις προς τις φορολογικές αρχές. Έχουμε λοιπόν και συμφωνίες αποφυγής της διπλής φορολόγησης με άλλες χώρες, πάνω από 30 συνολικά, οι οποίες προσαρμόστηκαν στους νέους νόμους. Άρα, οι ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται και όταν πρόκειται για περιπτώσεις φοροδιαφυγή, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την συμφωνία για τον φόρο στην πηγή, και αυτές είναι οι συμφωνίε που έχουν γίνει με την Ομοσπονδία Γερμανία και με τη Μεγάλη Βρετανία, εκεί η Ελβετία ασκεί μια στρατηγική του καθαρού χρήματο Οι δύο αυτέ συμφωνίε έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι δηλαδή πρόκειται αντίθετα με την, με την ε, τη συμφωνία για την φορολόγηση των τόκων που δεν είναι απελευθερωτικός τόκος είναι μια παρακράτηση του 35% εν αναμονή της φορολογίας, της φορολόγησης μάλλον που ελπίζουμε ότι θα γίνει εκ των υστέρων ο φόρος απελευθερωτικός φόρος στην πηγή ε, είναι οριστικός φόρος και καλύπτει κεφάλαια και μερίσματα, προσφέρει επομένως ευρύτερη φορολογική βάση από ε, την φορολόγηση των καταθέσεων. Και ο στόχος είναι να αποφευθεί ώστε ένας φορολογούμενος είτε χώρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε άλλης, όταν έχει καταθέσει την Ελβετία να αποφεύγει την φορολόγηση στην χώρα καταγωγής του. Γι' αυτό και τα ποσοστά είναι προσαρμοσμένα και με αυτά της χώρας ε, ε, προέλευσης. Με ρωτήσατε και για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται βέβαια να προβεί σε παρόμοια συμφωνία, σε παρόμοια συμφωνίας με την Ελβετία. Εμείς είπαμε ανέκαθεν ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε τις χώρες οι οποίες επιθυμούν να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να εξυπηρετήσουμε την φοροδιαφυγή ή την φοροαποφυγή από τις εθνικές φορολογικές αρχές. Αυτός ο φόρος που ανέφερα πριν θα είναι ένας, τρόπο τρόπος να λυθούν και τα προβλήματα του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος με μια συμβατότητα με την καταβολή φόρων και ταυτόχρονα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπέρ της οποίας δεσμεύεται η Ελβετία. Ίσως η πρόεδρος της ε, πολιτικής μας επιτροπής είναι διατεθειμένη να συμπληρώσει. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικώς χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων του σημερινού απογεύματος. Θα έρθω πολύ σύντομα στο ερώτημα πού υπάρχει περιθώριο για την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα πρώτα να τονίσω ότι η, πολιτική, η Επιτροπή μας Εξωτερικής Πολιτικής του Εθνικού μας Συμβουλίου ασχολείται πολύ ενεργά με την ευρωπαϊκή πολιτική που αποτελεί η συνεργασία μας δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολύ υψηλή προτεραιότητα. Εγώ βλέπω δύο δυνατότητες, καταρχήν για μια ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που όπως είπε και η πρόεδρός μας η οποία συνεργασία λοιπόν είναι ήδη πολύ στενή. Αφενός έχουμε ορισμένα οικονομικά εμπόδια λόγω του ότι η Ελβετία είναι τρίτη χώρα. Δεν είναι με μέλος της ενιαίας αγοράς, ούτε καν της Τελωνιακής Ενώσεως και έχει και δικό της νόμισμα. Έχουμε όμως πολύ, στενές εμπορικές, πολύ στενή εμπορική συνεργασία. 60% των εξαγωγών μας βαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και 80% των εισαγωγών μας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συμφωνήσει κάποιες, κάποια ανοίγματα τομεακά. Υπάρχουν και ορισμένοι τομείς όπου μπορούμε να προωθήσουμε ακόμη αμοιβαία το άνοιγμα. Αυτό προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το δικό μας, της Ελβετίας. Η δεύτερη δυνατότητα βελτίωσης και στενότερης συνεργασίας είναι πολιτική και θεσμική, όπως εξήγησε ήδη η Πρόεδρός μας. Συνεργαζόμαστε και στην εξωτερική πολιτική και σε περιπτώσεις, ας πούμε, περιοχών κρίσεων κλπ. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά, αλλά και στα πλαίσια διεθνών οργανισμών. Ιδιαίτερα με τον νέο ρόλο τον πλέον ενισχυμένο δημοκρατικό ρόλο που ε, μπορεί να ασκήσει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να εντείνουμε και τη συνεργασία μεταξύ ημών και του δικού μας Κοινοβουλίου. Έχουν ήδη αρχίσει, έχουν ήδη ε, εντατικότερες επαφές μεταξύ των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Ελβετικού Κοινοβουλίου. Αυτή η ανταλλαγή είναι πραγματικά σημαντική για να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση και να ενισχυθούν οι σχέσεις. Ξέχασα να απαντήσω στο ερώτημα για τη διαδικασία της κινητικότητας. Αποτελούμε μέρος του χώρου Σέγγεν και τη Συμφωνία του Δουβλίνου. Κατά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης, η Ελβετία τήρησε θέσεις που ήταν πολύ κοντινές με, τις με των περισσότερων κρατών μελών Δηλαδή δεν βρίσκεται καθόλου σε ακραία τοποθέτηση. Πολύ ωραία. Ο λόγος στον κύριο Ντανζάν, τον ε, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Κυρία Πρόεδρε, υπενθυμίσατε τον ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα σας σε μια σειρά από διαιτησίες και διαμεσολαβήσεις για τη διπλωματική σας ικανότητα που κατέβνασε κρίσεις, ε, σειράξεις, ε, αντιπαραθέσεις διάφορους ευρωπαϊκούς, ευρωπαϊκές περιοχές όπως τα Βαλκάνια. Για τον Νότιο Κάφκασο που είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή είχα δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς αποτιμάτε το ενδεχόμενο μεταξύ Ρώσων και Γεωργιανών να ξαναρχίσει ο διάλογος, κάτι που στο επίπεδο του ΟΗΕ της Γενέβης δεν φαίνεται πολύ πιθανό, και έπειτα η χώρα σας, ε, στην περίπτωση των Βαλκανίων, είδαμε να μπορεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ δύο ισχυρών ε, υποστηρικτών. Εσείς από άποψη μηχανικής τοποθέτησης, πώς θα μπορούσατε ε, να τοποθετηθείτε σε σχέση με την ευρωπαϊκή διπλωματία. Υπάρχει συγκεκριμένο διάβλο που μπορείτε να διαθέσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορείτε να στηρίξετε λόγω χάρη εμά ω μία από τι πλευρέ που στηρίζουμε κάποιου σε μια αντιπαράθεση. Ευχαριστούμε κύριε Ντανζάν, ο κύριος Λούνατσακ. Κυρία, Κυρία Λούνατσακ. Ευχαριστώ. Κυρία, κύριε Πρόεδρε, καλώ ορίσατε κυρία Καλμιρέη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα τελείωσαν τα γαλλικά όμω. θα σα μιλήσω γερμανικά προέρχομαι και εγώ από την γειτονική σας χώρα, από κύριο Σβόμποντα, την Αυστρία δηλαδή, και ως Αυστριακή αλλά και ως εκπρόσωπος των Πράσινων, θα, ε, εκφράσω, θα, θα εξέφραζα την χαρά μου εάν η Ελβετία γινόταν ε, μέλος, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατανοώ και πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο υπάρχουν μεταξύ των Ελβετών τόσο πολλοί που δεν θέλουν και να συμμετέχουν και στη λήψη των αποφάσεων και όχι μόνο στο να πληρώνουν. Αλλά παρόλα κυρία Πρόεδρε, λίγα σχόλια για τις εξωτερικές σχέσεις και μετά θα έρθω και στο τραπεζικό απόρριτο. Μίλησατε ήδη για τα Δυτικά Βαλκάνια και εγώ εδώ εκτιμώ πολύ την ε, συμμετοχή και τη συμβολή της ε, Ελβετίας, ιδίως στην Eulex, είμαι και εισηγήτρια για τη σχετική έκθεση, γνωρίζω ότι στην Ελβετία υπάρχει μεγάλη κοινότητα Αλβανών από το Κόσοβο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το γεγονός ότι δεν έχουν αναγνωρίσει όλες οι χώρες μέλη το Κόσοβο, ορισμένες και λόγω προβλημάτων με μειονότητες που έχουν ε, στις δικές τους επικράτειες. Μήπως <clears throat> θα μπορούσατε κι εσείς να τις παροτρύνετε και να τους εξηγήσετε ότι περισσότερη αναγνώριση για το Κόσοβο <clears throat> θα ήταν το σημείο όλη τη Ευρώπη Δεύτερο, Νότιο Κάφκασο, ο κ. Ντονζάν μίλησε σχετικά. Γνωρίζω το έργο τη, ε, κ. Ταλιαβίνη, τη Ελβετίδας ε, τεχνικού, ε, η οποία ασχολήθηκε με τα προκαταρκτικά στάδια των ένοπλων συγκρούσεων. Βλέποντας, εξετάζοντας δηλαδή πώς ανεβαίνουν οι τόνοι και το μίσος, έστω και φραστικά, στα προκαταρκτικά στάδια. Ε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς βλέπετε τις ε, συνομιλίες της Γενέβης και τις ενδεχόμενες πρόπτικες. Τώρα, για το τραπεζικό απόρριτο. Είπατε ότι η Ελβετία επιθυμεί να παίξει ρόλο πρωτοπόρου. Μιλήσατε για τον νόμο περί πλησίματος του βρώμικου χρήματος. Είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει να έχετε στις τράπεζες σας χρήματα από φοροφυγάδες στις πατρίδες τους. Το γεγονός όμως, ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, και εμείς ακούσαμε από ε, κύκλους της ελληνικής κυβερνήσεως ότι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ από ελληνικές περιουσίες έχουν κατατεθεί σε ελληνικές τράπεζες που επομένως δεν φορολογήθηκαν στην Ελλάδα. Είπατε οι, ίδιες, είπατε η ίδια ότι ενδέχεται να προχωρήσετε στη σύναψη μιας ειδική συμφωνίας με την Ελλάδα και η Ελλάδα φαντάζομαι είναι σύμφωνη. Αλλά ίσως αυτό θα πάρει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Εν ώψη αυτής της δραματικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε τώρα στη χώρα αυτή, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο και πριν να υπάρχει αυτή η συμφωνία να δοθούν κάποιες δυνατότητες στα χρήματα αυτά τα οποία πιθανώς και ε, ε, πολύ πιθανώ βρίσκονται σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ε, ως προϊόν φοροδιαφυγή, να διατεθούν σε ελληνικές αρχές και να μην παραμείνουν απλώ σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κύριε Λούνατσεκ, ο κύριος Ρούμπιχ, αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσει μας με την Ελβετία. Ευχαριστώ. ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημερινή συνάντηση. Δηλώνω ότι κολλείεται και ο Γκάλαχερ. Στα πλαίσια των από μακρού χρόνου σχέσεων μας με τα 26 της Καντόνια και τις τρεις γλώσσες της η Ελβετία έχει αποτελέσει για πολλά χρόνια και το πρότυπο για την Ευρώπη που καταφέρνει και συνεργάζεται θαυμάσια και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 χώρες μέλη και 23 ε, γλώσσες. Έχουμε μάθει πολλά από την Ελβετία λοιπόν και στο μέλλον είμαι βέβαιος θα μάθουμε επίσης πολλά πράγματα, για παράδειγμα στον τομέα του φόρου προσθεμένης αξίας που το σύστημα, το σύστημα το δικό σας είναι πολύ προοδευτικό και σύγχρονο και όπου θα μπορούσε από αυτό να υποφεληθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή επίσης ε, η προσπάθεια εξυγίανσης της τράπεζας UBS που θα έπρεπε και από εκεί να διδαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και άλλα σχετικά θέματα. Θα, ζητήσω, θα σας ευχαριστήσω μάλλον και για τον τομέα της ενέργειας που διατηρήσατε ανοιχτές τις επαφές με το Ιράν και ιδίω με τις θετικές δυνάμεις του Ιράν και παίξατε έναν ουδέτερο διαμεσολαβητικό ρόλο, διότι βεβαίως συνολικές κρίσεις δεν είναι ε, πάντοτε οι πιο χρήσιμες. και αφήνοντας θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων απ' έξω. Θα ήταν σημαντικό και για τον τομέα της ενέργειας να συμμετάσχει η Ελβετία στον Ευρωπαίο Ρεθμιστή Ενέργειας, ΕΣΑ, διότι οι αγωγοί που θα διέρχονται την Ευρώπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δυνατότητες αποθήκευσης στην Ελβετία είναι ασφαλώς σημαντικό κίνητρο ώστε να μπορέσουμε να διταχθούμε και σε αυτούς που ζητούν τη διατήρηση των πυρηνικών σταθμών, αλλά και διεθνώς θα ήταν σκόπιμο να κάνει σχετικά βήματα η ε, Ελβετία στο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Εδώ η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία έχει διεξαγάγει πολλές συζητήσεις και χαιρόμαστε διότι σήμερα καθίσταται δυνατόν να συνομιλήσουμε και μαζί σας και ευχόμαστε να ενταθεί και να γίνει ακόμα πιο στενή η συνεργασία μας με την Ελβετία και στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Ρούμπι, ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Καλμίρεϊ. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος που συμπαρασταθήκατε και στην Task Force ε, στην ε, την Ινησία. Εγώ μπόρεσα να μεταβώ στη, στο πλευρό της κυρίας Άστον στην επίσκεψη αυτή και ευχαριστώ ιδιαίτερα στη χώρα σας για τη συμβολή της σε θέματα όπως και η λεύκανση παράνομων προσόδων και γενικότερα σε ό,τι οι ανάγκες υπήρξαν στην Τινησία. Ήσασταν πραγματικά πολύ επικοδομητικοί. Με συγχωρείτε που έφτασα κάπως αργά, είχα άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όμως μπορεί να πει κανείς ότι η Ελβετία είναι ένας σημαντικός εταίρος μας σε ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως τα ζητήματα του δημόσιου χρέους, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ε, οργανωμένη εγκληματικότητα, δυσκολίες και διενέξεις όπως αυτή με, την, ε, με τα προβλήματα της Κολομβίας, όπου ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση. Γενικώ είναι πολύ ενεργό ο ρόλος της Ελβετίας στην καταπολέμηση της θερμοκρατίας. Αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων ταυτόχρονα. Έχετε λοιπόν ε, έναν παραδοσιακό ρόλο που έχετε αναλάβει εδώ και σε θέματα της ασφάλειας Τη ενεργειακή διαφοροποίηση, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. ω μέλο λοιπόν του χώρου Σέγγεν έχετε παρόμοια προβλήματα όπω και εμεί λόγω χάρη αυτών των δημογραφικών εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ήδη κάποιε προβλέψει για την ερχόμενη 35 ετία. Οπότε τώρα εντό εισαγωγικών σε ένα πιο αθλητικό πνεύμα θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφιλειωθούμε με ορισμένες ε, θέσεις που μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας ε, εθνικές θέσεις. Και το λέω αυτό με μεγάλη μετριοπάθεια καθώς χάσαμε τις εκλογές. Όμως ουσιαστικά κέρδισε ο Ελβετός υποψήφιος υπουργών εξωτερικών Χάσαμε εμείς και νικήσατε εσείς. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις προσπάθειές σας και την ε, προσφορά σας στην ε, στήριξη της Τινησίας. Ήταν πολύ σοβαρή η συμβολή σα σε όλες αυτέ τι περιπτώσει. Σα ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Κλείνει η συζήτηση με τον κύριο Σφαμπ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως. Ευχαριστώ για την επίσκεψή της, την Πρόεδρο κυρία Καλμιρέη, με την έλευσή σας εδώ δείχνετε ότι εκτιμάτε και εσείς το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ανδρώνεται μέσα στην, στον ρόλο του, του πλήρου συνομοθέτου. Ίσως η Επιτροπή Εξωτερικών είναι υπερβολικά πολιτικοποιημένη για να συζητήσει ορισμένα θέματα τα οποία α, τίθενται στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των, α, της, Ελβετίας και των χωρών της Ένωσης. Γι' αυτό και πολύ θα χαρώ να ξαναέλθετε, κυρία Πρόεδρε, και να επισκεφθείτε και άλλες επιτροπέ επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα επανέλθω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς. Εγώ βρίσκω ότι αυτό ως δήλωση είναι τολμηρό. Αν εξετάσουμε τις οικονομικές εξελίξεις μπορούμε να διατυπώσουμε καθαρά την ε, θέση ότι είστε από τους πλέον ενεργούς εταίρους και ελπίζω μάλιστα αυτό να ενισχυθεί και στο μέλλον. Από αυτό προκύπτουν βέβαια και πολιτικές υποχρώσεις που δεν είναι πάντοτε εύκολο να τις επομιστεί η κυβέρνησή σας μέσα στο σύστημά σας άμεσης δημοκρατίας με τις ε, διάφορες δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται, αλλά θα ήταν ασφαλώς εσφαλμένο να προκαλείται η εντύπωση ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της ενιαίας αγοράς. Το αντίθετο ισχύει. Το αντίθετο είναι καλό και το αντίθετο πρέπει να ε, γίνει σαφές και στους συμπολίτες σας. Και πολύ θα ήθελα αυτό το μήνυμα να το μεταφέρετε. Ευχαριστούμε κύριε Σφαμπ. Ας αφήσουμε λοιπόν πολύ χρόνο στην Πρόεδρο για να απαντήσει στα πολύ άριθμα ερωτήματα που ακούσαμε. Παρακαλούμε. Θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας για την ειρήνη και τις προσπάθειές μας για διαμεσολάβηση και διτησία. Εδώ άκουσα για την θετική αποτίμηση των προσπαθειών μας στις σχέσεις Ρωσίας-Γεωργίας. Ε, πρέπει να σας πω ότι πράγματι είμαστε διαμεσολαβητές, ενεργούμε κατά τρόπο όσο το δυνατόν αντικειμενικό μεταξύ δύο πλευρών και είμαστε διάμεση και στη διαδικασία προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Δεν πρόκειται για απλό ζήτημα, διότι αναζητούμε ένα σύστημα ελέγχου και διακόμισης των εμποραυμάτων σε ουδέτερες συνθήκες Καταλαβαίνετε όμως τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει με την ε, Οσετία και την ε, Αμπχαζία σε αυτό το πλαίσιο. Καταλαβαίνω λοιπόν από το βαθμό δυσκολίας του ρόλου μας ως διαμεσολαβητών που είναι σοβαρότατες οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε οι δύο πλευρές είναι αρκετά συναισθηματικές στην περίπτωση αυτή, πόσο σημαντική είναι η διαμεσολάβησή μας. Αυτή μας ζητήθηκε από τις δύο ακριβώς πλευρές. Δεν παρεμβαίνουμε ουδέποτε χωρίς αίτημα από πλευράς των δύο μερών που μπορεί να έχουν κάποια διαφωνία. Πρέπει να έχουμε τη δική τους συνένεση, τη δική τους συμφωνή γνώμη. Δεν Μάλλον γνωρίζω καλά και τις δύο πλευρές, αλλά δεν θα σχολιάσω καμία πολιτική θέση, ούτε θα λάβω καμιά πολιτική απόχρωση, διότι πρέπει να είμαι ουδέτερη ως διαμεσολαβήτρια. Ελπίζω απλώς ε, να είναι ικανοποιητικέ οι λύσεις που θα προτείνουμε ε, και για τους μεν και για τους δε, αν και ίδιων όλων των συμβιβαστικών λύσεων να μην ικανοποιούν απόλυτα ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Θα κάνουμε πάντως ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σε αυτές τις προσπάθειες διαμεσολάβησης δεν έχουμε συγκεκριμένη σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτω ή άλλω δρούμε κατόπιν αιτήματο των δύο πλευρών. Δεν ελήφθη τέτοιο αίτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από την Γεωργία. Εργαζόμαστε λοιπόν ε, με την πρόσκληση των δύο πλευρών, όμως ε, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους διεθνείς παράγοντες του διεθνούς προσκυνείου ε, ε, στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς προχωρούν οι εργασίες μας. Το ίδιο και για τις διαπραγματεύσεις μας με τη Ρωσία στα εμπορικά ζητήματα, προκειμένου η Ρωσία, η Ρωσία να προσχωρήσει στον ΠΟΕ τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύει το ίδιο όπως την διαμεσολάβησή μας για την Αρμενία και την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους αλλά ενημερωτική. Οπότε εκεί να πούμε ότι όχι, να πούμε μάλλον ότι δεν δρούμε κατόπιν εντολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κατόπιν αιτήματο των δύο πλευρών που μπορεί να ανακύψουν. Τώρα, για το θέμα του Κωσυφοπεδίου και των Βαλκανίων εμείς ε, συμμετέχουμε στην Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο, στην ε, Καφόρ, καθότι είναι μια από τις λίγες χώρες από η Ελβετία δραστηριοποιεί το στρατό της. Ε, είμαστε πολύ, φιδόμαστε ιδιαίτερα της παρουσίας των στρατιωτών μας σε ξένες επικράτειες, αλλά στο Κωσυφοπαίδιο συμμετέχουμε με 200 περίπου, με 200 περίπου άντρες. Επίσης στη Γιουφόρ στην Βοσνία με ένα εσωτερικό τάγμα πολύ πιο περιορισμένο. Και εκεί συμμετέχουμε. Για μας το κοσυφοπαίδιο είναι σημαντικό, σωστά το τονίσατε κυρία μου, επειδή υπάρχει σημαντική κοινότητα κοσοβάρων στην ε, Ελβετία. Υπήρξαμε οι πρώτοι που προωθήσαμε το σύνθημα status before standards, δηλαδή για, αν δεν γίνουν ε, πρόοδοι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την της δημοκρατίας, μόνον εφόσον έχει προϋπάρξει η αναγνώριση του καθεστώτος της χώρας θα το πετύχουν αυτό οι πολίτες. Έτσι λοιπόν, ίσως οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του κοσφοπεδίου να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με το δικά μα, όμω υπάρχει πλέον ένας συνομιλητής ένας συνομιλητή που έχει υπόσταση και με τον οποίο μπορούμε και εμείς να συνομιλούμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία μας στη χώρα αυτή είναι διαρκή και αυτό είναι πολύ προτιμότερο από την ασάφεια που επικρατούσε προηγουμένω. Ω προ το τραπεζικό απόρριτο, κυρία μου, τα 200 δι έφυγαν από την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήρθαν στην Ελβετία. Υπερτιμούμε κάποιε φορέ το τι έχουμε στα χρηματοκιβατιά μα στην Ελβετία. Σα διαβεβαιώ, τα χρήματα αυτά δεν βρίσκονται όλα στα ελβετικά θησαυροφυλάκια. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Ελλάδα που έδειξε ενδιαφέρον για έναν φόρο στην πηγή και βάσει αυτού του προτύπου συνάψαμε και δύο παρόμοιες συμφωνίες με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έναυσμα για τις συζητήσεις μας με άλλες χώρες. Όχι μόνο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους μπορεί να ενδιαφέρουν. να ενδιαφέρει μάλλον η θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Για τη διαδικασία της ένταξης Πολύ σωστά είπατε κύριε Ρούμπιχ ότι αυτή η διαδικασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια διαδικασία ένταξης που διαρκεί περίπου 720 χρόνια και οδήγησε στην ίδρυση της Ελβετίας με καντόνια, τα οποία ήταν κυρίαρχα κράτη τον 12ο αιώνα με το δικό τους νόμισμα. Το, πρώτο, το δικό μας ελβετικό νόμισμα έχει ηλικία 150 ετών περίπου. Σιγά σιγά λοιπόν τα καντόνια αυτά χώρισαν εξουσίες στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένα πρότυπο ενταξιακό το διαθέτουμε και εμείς από μόνοι μας. Ξέρουμε λοιπόν πώς ε, προχωράει η ένταξη στην ε, Ευρώπη. Άλλωστε σύστημα εναλλαγής των προεδριών ε, υπήρχε και σε εμά σύστημα που μπορεί να παρομοι... παρομοιαστεί με το δικό σας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης, ό,τι αφορά την ενέργεια, στον τομέα της ενέργειας, Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία για την ηλεκτρική ενέργεια, ιδίω για την ε, μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια προ τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τη σταθερότητα παροχή ηλεκτρισμού. Εμεί είμαστε μια χώρα διέλευση μεταξύ βορρά και νότου τη Ευρώπη για την ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε για άλλη μια φορά βλέπουμε η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν κοινά συμφέροντα για τη σύναψη μια τέτοια συμφωνία. Βεβαίω, ε, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η σύναψη μιας τέτοια συμφωνία ε, παρακολύεται ελαφρώς, καθυστερεί, ε, λόγω θεσμικών προβλημάτων. Κάποιος ανέφερε, νομίζω κύριε Σφάπ εσείς, ότι η Ελβετία δεν είναι μέρος της εσωτερικής αγοράς. Ναι, δεν είναι. Έχει όμω τομεακή πρόσβαση στην ε, αγορά η Ελβετία. Δηλαδή έχει πρόσβαση στου τομεί που καλύπτονται από κάποιε συμφωνίε. Αλλά όχι κατά τρόπο γενικευμένο. Ε, από τις διμερείς συμφωνιε τι τομεακέ διμερείς συμφωνιε που κατά καιρού έχουν συναυθεί. Οπότε εταιρικέ σχέσει υπάρχουν μόνο εκεί. Λόγου χάρη. Υπάρχει εταιρική σχέση για τα ζητήματα τα φορολογικά ε, για τα ζητήματα που αφορούν τη φορολόγηση τη αποταμίευση. ή το ίδιο για την μετανάστευση, αυτά που καλύπτονται από τη Συμφωνία του Δουβλίνου ή την πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένου τομεί τη γεωργικής αγορά. Εκεί έχουμε πρόσβαση και σε περιπτώσεις που καλύπτονται από συμφωνίες. Γενική πρόσβαση δεν υπάρχει. Δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διμερής, λοιπόν, ο διμερής διάβλος καθιστά απίθανε την προοπτική να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου προκειμένου να έχουμε γενικευμένη πρόσβαση στην αγορά, την ενία. Αλλά θεσμικά ζητήματα υπάρχουν και στην Ελβετία. Δηλαδή θα έπρεπε να πλουστεύσουμε τις σχέσεις μας που έχουν γίνουν εξαιρετικά περίπλοκες ε, εξαιτία των μεικτών επιτροπών, των υποεπιτροπών, των ομάδων εργασίας που δημιουργούνται. Ο κίνδυνος είναι να σκοντάφτει κάθε φορά ο κίνδυνο στο πώ θα υλοποιούνται και θα εφαρμόζονται οι διμερεί συμφωνίε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε διερευνητικέ συζητήσει για τα θεσμικά ζητήματα που μα απασχολούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Μπαρόζο και εγώ η ίδια συζητήσαμε για το ενδεχόμενο κοινή και συντονισμένη προσέγγισης Δηλαδή, τα ζητήματα ενδιαφέροντο και για τι δύο πλευρέ βρίσκονται επιτάπητο συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών ζητημάτων. Η διαπραγμάτευση θα υπάρξει στα πλαίσια ενό κοινού πακέτου, ένα τρίτο πακέτο διαπραγματεύσεων διμερών με την Ελβετία. Να το ξαναπώ, για την Ελβετία αυτό θα είναι το μέσο να έχουμε μια εταιρική σχέση πρωτίστη σημασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε ο πρώτος ε, εταίρο μας από άποψη οικονομικής και πολιτικής. Θέλουμε λοιπόν η εταιρική σχέση αυτή να ενισχυθεί. Το status quo δεν είναι λύση, πρέπει να ενδυναμωθεί, να ε, ενεργοποιηθεί αυτός ο διμερή διάβλο και αυτό θα γίνει μέσα από διαπραγματεύσει που απλέ δεν θα είναι ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για την Ελβετία. Έχουμε όμως όλη την καλή θέληση να είμαστε επικοδομητικοί σε αυτή την εταιρική μας σχέση. Ως προς τα προβλήματα γειτονία που αναφέρθηκαν είναι προφανές. Υπάρχουν μεταξύ γειτόνων προβλήματα γειτονία. Υπάρχουν όμως και αρμόδιες ομάδες εργασίας που αναζητούν πρακτικές λύσεις στα προβλήματα γειτονία. Υπάρχουν τριμερείς ομάδες εργασίας Οπότε νομίζω τα ζητήματα των εγγυήσεων και ούτω καθεξής θα εξεύρουν λύση. Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζουμε και εμείς τα ίδια προβλήματα στις σχέσεις, στις μας με τις όμορες χώρες. Και μάλιστα πολλέ φορέ η δυσκολία μα είναι μεγαλύτερη να ενεργήσουμε στην Ιταλία και την Γαλλία και την επικράτειά του λόγω κάποιων δυσκολιών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Πρέπει λοιπόν και στι μεν και στι δε περιπτώσει να βρεθούν λύσει όπως για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η Ελβετία δέχτηκε με δημοψήφισμα την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Εάν την αποδεχτήκαμε λοιπόν την συμφωνία αυτή με συνοδευτικά μέτρα τα οποία στόχο έχουν να εξασφαλίσουν στους πολίτες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται στην Ελβετία τις ίδιες μισθολογικές συνθήκες και τις ίδιες συνθήκες εργασίας όπως αυτές που ισχύουν για τους Ελβετούς, για να μην υπάρχει εργασιακό ντάμπινγκ, παρόλα αυτά δυσκολίες απομένουν. Όπως και μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση της Ελβετίας όμως είναι ιδιαίτερη ιδιάζουσα θα έλεγα, διότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών που έρχονται να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην ε, Ελβετία. Το 2008 είχαμε 4.000 Γερμανούς το μήνα που έρχονταν στην περιοχή της ε, Ζηρίχης και σήμερα 250.000 άτομα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταφτάνουν κάθε πρωί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εργαστούν στην Ελβετία. Είμαστε ορθάνυχτοι. Όμως ε, για τα συνοδευτικά μέτρα που έγιναν αποδεκτά την ίδια στιγμή με τη Συμφωνία της Ελεύθερης Κυκλοφορίας ε, των Προσώπων από τον ελβετικό λαό, τα συνδευτικά αυτά μέτρα είναι πολύ σημαντικά για, την, ε, για το κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό το εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό που τόσο χρειαζόμαστε, αλλά που κάποιες φορές κάποιους τους ε, ενοχλεί. Θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ανταγωνισμό σε σχέση με το τοπικό εργατικό δυναμικό. Δεν είμαστε λοιπόν οι μόνοι που αντιμετωπίζουμε τέτοιου προβλήματα. Η Ελβετία, συγγνώμη, είναι πάντοτε επικοδομητική όμως στην αναζήτηση λύσεων. Συζητήσαμε μεταξύ Ελβετία και Γερμανή. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και είμαι βέβαιο ότι θα βρούμε μέτρα να εφαρμόσουμε απόλυτα πρακτικά και ικανοποιητικά για όλου. Ίσως θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι η συνάδελφο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για την Ελβετία ε, οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι ταυτόσιμες ε, και γι' αυτό στον τομέα της εξωτερικής ε, πολιτικής είναι προσυμφέρον όλοι να συνεργαστούμε για να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Δείτε τι συμβαίνει στα Βαλκάνια, στη Αφρική, στον Κάφκασο. Πρόκειται για πολύ σοβαρά προβλήματα και μην ξεχνάτε ότι δεν μοιραζόμαστε μόνο μία κοινή γεωγραφική θέση ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή, αλλά ένα κοινό πολιτισμό κοινέ γλώσσες και επίσης ε, είμαστε και εμείς υπέρ της πολιτιστικής πολυμορφίας την οποία υπερασπίζεται και η Ελβετία. Ε, αυτή είναι η βάση των στενών σχέσεων ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 20 χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, της αρχής της δεκαετίας του 90, αντιμετώπισε και η Ελβετία μια κρίση χρέους λόγω μιας κερδοσκοπικής φούσκας ενυποθήκων δανείων πλέον ε, και χρειάστηκε το κράτος να διασώσει μια σειρά από τράπεζες αυτό οδήγησε σε ένα πάρα πολύ υψηλό ε, δημόσιο χρέος και χρειάστηκε να βρούμε και εμείς σε μία λύση. Τελικά καταφέραμε να θέσουμε υπό έλεγχο το πρόβλημα αυτό υιοθετώντα ε, διάφορα οικονομικά μέτρα και θεσπίζοντα ε, και ένα νέο μέσο, το φρένο για το δημόσιο χρέο ε, που εγκρίθηκε κατόπιν δημοψηφίσματο. Ούτω ώστε να μην μπορεί μία γενιά να δαπανίσει όλο το κληροδότημα της χώρας μας και έτσι διαφυλάττουμε τις μελλοντικές γενναίες. Ε, οπότε έτσι αποφεύγουμε τα ε, ε, πολύ ψηλά δημόσια χρέη και κάνουμε χρηστή διαχείριση των δημοσιοοικονομικών μας. Ε, σήμερα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα δημοσίου χρέους και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να ανταλλάξουμε απόψεις. Κύριε Σοβάμπ, Είπατε ότι δεν ανήκουμε στην εσωτερική αγορά. Ε, ε, ε, de facto όμως είμαστε τόσο στενά συνδεδεμένοι με αυτή την εσωτερική αγορά. Πάνω από ένα εκατομμύριο υπήκοοι ευρωπαϊκών κρατών διαβιούν στην Ελβετία και εκατομμύρια Ελβετοί μένουν, ε, ζουν ε, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι Ελβετοί καθημερινά πηγαίνουν να δουλέψουν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντίστροφο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και θα ήθελα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να συνεχίσουμε αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Μακπάρντερ. Εγώ θα ήθελα με αυτήν την ε, ε, θερμή ευχαριστία να εκφράσω την ευχαρι... τις ευχαριστήσεις μου και προς τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Απλώς να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που μόλις άκουσα από την κυρία Μακβάλτερ και ως προς τα σχόλια του κυρίου Σφάμπ. Σήμερα συμπληρώσαμε τις συζητήσεις που ήδη γίνονται σε διάφορες επιτροπές και προσχολούνται με πιο λεπτομερείς συγκεκριμένα ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος μεταφορές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, περιβάλλον και το καθεξής. Πιστέψαμε ότι Συνενώντα σήμερα όλε αυτέ τι πτυχέ, γιατί είναι πολύμορφο αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται μπροστά μα, ε, σχολιάζουμε ουσιαστικά την εξωτερική μα πολιτική. Δεν μιλάμε για μία μόνο πτυχή μια από αυτέ τι διμερεί συμφωνίε. Σκοπό τη συνάντησή μα ή ο σκοπός μάλλον της συνάντησής μας πιστοποιείται και από το γεγονός ότι κατά την επίσκεψη του Προέδρου μας Μπούζεκ στην Ελβετία Μαζί του μετέβησαν και πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με συγκεκριμένε πτυχέ διαφορετικών συμφωνιών. Υπάρχει παρόλα αυτά ένα γενικότερο τοπίο το οποίο νομίζω ότι άξιζε την προσοχή τη Επιτροπή μα και των μελών τη. Σα ευχαριστούμε λοιπόν για την προσέλευσή σα. Καλή δουλειά για όσα έχετε ακόμη να κάνετε σήμερα και καλή επιστροφή στη χώρα σας. Ίσως η επόμενη συνάντηση σύντομα να οργανωθεί στη δική σας χώρα. Ε, abbiamo ε, minuti di attesa perché... Έχουμε 10 λεπτά κενό. Οι ψηφοφορίε πρέπει να αρχίσουν ακριβώ ε, βάσει του προγράμματο στι 4.30. Οπότε διακόπτουμε για 10 λεπτά. όπως σωστά με τα νεύματά του επιβεβαιώνει ο συνάδελφος, ο αγαπητός φίλος κ. Άτκινς. Λοιπόν, στις 4.30 θα ξαναρχίσουμε. Bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo... Είναι 4.30 συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Ωστόσο, θα σας παρακαλούσα να είχατε την ευγενή καλοσύνη να μου επιτρέψετε να αλλάξουμε τη σειρά των ψηφοφοριών, διότι η συνάδελφος Μακόπη δεν είναι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, έχει συμμετοχή σε άλλη επιτροπή. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε με μια από τις υπόλοιπες εκθέσεις, την τελευταία τι ψηφοφορίε και να ψηφίσουμε την πρώτη μόλις έρθει η συνάδελφος Μακοβέη. Φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση, οπότε εάν συμφωνείτε θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, αντιμετωπίζοντα τι προκλήσει και ξεπερνώντα τι δυσκολίε. Ελπίζω να συμφωνεί και ο εισηγητή, ο κ. Κράισλ Ντέρφλερ. Αν έχετε λοιπόν τι κάρτε τη ψηφοφορία, περνάμε στην ε, τροπολογία 63, καθότι 62 αποσύρθηκε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Καλύτερα να ελέγξουμε και ηλεκτρονικώς. Για την 68 άρχεται η ψηφοφορία. 68. Πέρας. Ξεκάθαρο, 21 προς 14 εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απορρίπτονται οι 70 και 71, 72. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ε, αποσύρονται οι 73 και 74. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά ωστόσο για την 72 εντωμεταξύ. 72 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάποιοι ψηφίζουν χωρίς να βάζουν την κάρτα στο μηχάνημα, αλλά πρέπει να κλείσουμε την πληροφορία. 22 προς 16. Σαφώς απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. 77. 77. Ηλεκτρονικός έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 προς 19. 78 με την πρώτη προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αποσύρεται η 79-80. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86, τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Με συγχωρείτε. 3. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ κατά, αποχές, μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά θα ήθελα να το ελέγξω. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23 όχι και 22 ναι. Άρα απορρίπτεται. 95 με την προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 με προφορική τροπολογία την τρίτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100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 Αποχέ εγκρίνεται. Αποσύρονται 115, 116 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 και 118 παρομοιότυπε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 επέρ. κατά αποχέ. εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. 122 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. έναρξη της ψηφοφορίας. Καμιά φορά ακόμη και ο Όμηρος κοιμάται. Πέρας. 35 προς 21 απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120, 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 και 33 ε, παρομοιότυπες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεν είμαστε βεβαίοι, ναι, ε, με δύο μάτια και δυο ζευγάρια μάτια, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 132-33. Ε, μπορεί να συμβεί και αυτό. Πέρας. Πράγματι εγκρίνεται. 31 προς 26. Δύο ζευγάρια μάτια είναι πάντα καλύτερα. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην συμβιβαστική 10 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά θα προτιμούσα να το επιβεβαιώσω. 156 άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Πέρας.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 Κατά. Δεν είμαι βεβαίω Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. 171 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 προς 31 περνάει με δύο ψηφούς διαφορά. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά, αποχέ απορρίπτεται. 192 με προφορική τροπολογία, την 7η, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193 και 194 υπέρ, κατά, αποχέ. θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, αυτό το έλεγχο σίγουρα. Να το ελέγξουμε λοιπόν το 195. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 195. Πέρας. 26 προς 34 εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Ε, δεν το σηκώσατε το χέρι σας. Όμως Σα παρακαλώ να σηκώνετε κανονικά τα χέρια σα, γιατί τέλο πάντων θα περάσω 200. 200 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 202. Θέλετε πάλι έλεγχο. 201, εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη τη ψηφοφορία για τη 201. Πέρας. 31 προς 28 απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205, 211 συγγνώμη, 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 212 λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικός. Ε, όταν αμφιβάλλω, καλά κάνετε και με πιέζετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν, 212. Ε, μου φάνηκε ότι εγκρίνεται, αλλά πέρας. Μικρή διαφορά. 31 προς 29. Εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κανείς δεν εγκρίνεται 216. Α, λοιπόν. Κατά. Αποχές. Αυτή απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 220 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. 221 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Διασκεδάσατε. Πέρας. 28 προς 34 εγκρίνεται. Ε, παρόλα αυτά εγκρίνεται. Παρά την προπαγάνδα του κομματός μου. 1 και δύο. υπέρ. Κατά. Ε, δεν σηκώνετε πάλι τα χέρια. Πάλι θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ένα και δύο. Βαρεθήκατε λίγο, ε. Άρχεται η ψηφοφορία. 1-2. ενα Ένα-δύο. Ένα καθετος 2. Ε, μετά να σηκώνετε κανονικά τα χέρια, αλλιώς συνεχώς θα χάνουμε χρόνο. Πέρας τη ψηφοφορία. Επίτηδες το κάνατε. 61 προς 1. Με δουλεύετε. Θα αλλάξω γυαλιά. Τρία. Τροπολογία τρίτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6-7-8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11, 13 συγγνώμη. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά Αποχέ. Δεν είναι γιατί Γιατί 15 ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη τη προφορίας. Πέρας. 26 προς 36 εγκρίθηκε. 16. Παρακαλώ, κύριε Βότσον. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη του ΕΛΚ είναι στην αίθουσα και ψηφίζουν και πόσοι έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν. Μήπως ψηφίζουν περισσότεροι από όσου πραγματικά έχουν δικαίωμα. Το μηχάνημα, το ηλεκτρονικό τέλο πάντων μηχάνημα είναι σε θέση αμέσως να σας δώσει την πληροφορία που ζητάτε. Ε, ελπίζω τα μηχανήματα να λειτουργούν. Αυτόματο θα έπρεπε να είναι, για την ώρα δεν έχει φανεί να υπάρχουν ε, παρατυπίες. Πάμε στην 17. 17 υπέρ, κατά. Κατά για την 17. Απορρίπτεται. Την 16 τελικά δεν την ψηφίσαμε. Ας ψηφίσουμε για την 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη, 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 29-30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμμεμπαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 τροπολόγια 34 υπέρ, κατά, μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά θα προτιμούσα να ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 34. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 προς 28. 35-36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44, 44 υπέρ, κατά, δεν είναι ξεκάθαρο. 44, άρχεται η ψηφοφορία για την 44. Πέρας, 31 προς 31, γι' αυτό δεν ήταν σαφές, έτσι, ε, απορρίπτεται. 21, συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. 57. Εντάξει λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. 57. Πέρας. 30 προς 31. Τι να κάνουμε, εγκρίθηκε. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε αυτό. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa Πέρας. 24 προς 37 εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες της την γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. Παράγραφος πρώτη. Όχι, παράγραφος 6. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Μάλλον 10. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη β υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη σ υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη. Όχι, καλύπτονται όλα από την Επιτροπή Ανάπτυξη και έχουμε την τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 61 προς 1. Θρίαμβος. Θρίαμβος για τον εισηγητή. Bene, allora abbiamo, Έχουμε την Περιφερειακή Σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής. Τελική ψηφοφορία μόνον. Άρχεται ψηφοφορία. Δεν υπάρχει συγκητή στην αίθουσα, αλλά δεν είναι και τίποτα που μένει να συζητηθεί. Αβάντι, είναι πάμε. Γνώμη, δω, έκθεση παιδιό. Ας, ας μην έχουν έρθει. Δεν θέλετε να ψηφίσετε. Πέραστε τη ψηφοφορία. 50 προς 3. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία. Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αυστραλία για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από του αερομεταφορεί δεδομένων από τι καταστάσει επιβατών προ την υπηρεσία τελωνίων και προστασία των συνόρων τη Αυστραλία. Η κυρία Μακοβέη, συγγήτρια. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. 51-8, complimenti προς 8. Αγκρίνεται. Τώρα, Προεδρία, στον ευγενέστερο των αντιπρόεδρων μας, Πάσκο, καλό, καλή τύχη. Okay, let's uh, move along. Ας προχωρήσουμε. I would like those who, who have some other business. Ε, όσοι έχουν άλλες δουλειές και πρέπει να φύγουν, παρακαλούν να αποχωρήσουν. Ε, τώρα θα περάσουμε στις συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης, την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ Γεωργίας. Ε, κύριε Κρίστοφ Λίσε και στο εισηγητή, παρακαλώ, σα ακούμε. Szanowne Panie i Panowie Posłowie, e, nie chcę zabierać Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Δεν θα ε, καταναλώσω πολύ από τον πολύτιμο χρόνο σα Με μεγάλη ικανοποίηση δηλώνω ότι μόνο 59 τροπολογίες κατατέθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις οι τροπολογίες είναι ταυτόσιμες ή έχουν ίδιο περιεχόμενο και για το λόγο αυτό νομίζω ότι θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και στον χρόνο αυτό θα μπορέσουμε να εκπονήσουμε ε, το σχέδιο. Ευχαριστώ όλες και όλους τους και όλες για τη συνεργασία και θα ήθελα να προσθέσω ότι οι τροπολογίες δεν τροποποιούν θεμελιωδώς το μήνυμα του ψηφίσματος. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που ίσως μάλιστα υπερβαίνουν εν μέρη το αρχικό περιεχόμενο της συστάσεώς μου και ιδίως ιδίως σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των μεταρρυθμίσεων των αγώνα κατά της διαφθοράς. Έτσι λοιπόν οι τροπολογίες βαίνουν λίγο μακρύτερα από την αρχική μου πρόταση Εκφράζω την ικανοποίησή μου επίσης για το γεγονό ότι όταν μιλούμε για την γεωργία μιλούμε βέβαια την περίπλοκη θέση της χώρας αυτής με την, στην πράξη κατοχή μερών του, εδαφού, του εδάφους της, Απχαζία και Οσετία. Οι δύο αυτές περιοχές τελούν υποκατοχή, καθώς επίσης τίθεται και ορισμένα πολιτικά θέματα. Η αναγνώριση της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας από την Ρωσία ως ανεξάρτητων κρατών, ανεξάρτητων χωρών. Είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα που περιπλέκει την κατάσταση. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες. Η πλειοψηφία των τροπολογιών δεν αμφισβητούν, όπως είπα, το θεμελιώδες περιεχόμενο της ε, συστάσεως και υπάρχουν και ορισμένες τροπολογίες που όπως η ε, τροπολογία Φαγιόν από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Βεβαίω υπάρχουν ορισμένε ελλείψεις Σημαίνονται ορισμένε ελλείψει ε, στο κρατικό δόμημα της Γεωργίας, για παράδειγμα στην δικαιοσύνη, η πρόσβαση σε πληροφορίες. Αλλά βλέπω την δυνατότητα να εκπονηθεί συμβιβασμός και γι' αυτό προτείνω να συνεργαστώ, προσφέρω τη συνεργασία μου δηλαδή σε όλους τους κοιοδησίγητες, καθώς και στους συντάκτες και συντάκτριες τροπολογιών για να συζητήσουμε το περιεχόμενο των τροπολογιών τους και είμαι εν τέλει πεπισμένος ότι θα βρεθούν επαρκείς συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Πάσκου, η κ. Φαγιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, κύριο Λίσεκ, τον οποίο συγχαίρω επίσης για την έκθεσή του. Ο αριθμός των τροπολογιών, 59, δεν είναι υψηλός. Ίσως μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες και είμαι και διατεθειμένη βέβαια να συνεχίσω να διαπραγματεύομαι μαζί του για να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις η έκθεση τονίζει τις ε, σημαντικές προόδους της Γεωργίας καθώς και οι τροπολογίες εκείνες οι οποίες είναι κάπως επικριτικότερες δεν δείχνουν ότι είμαστε κατά της Γεωργίας αλλά θέλουμε απλώς να προσεγγίσει η χώρα αυτή ακόμη περισσότερο στις ευρωπαϊκές αξίες. συντάξει των τροπολογιών και εμείς τονίσαμε ότι πρέπει να ενταχθούν ξανά η Απχαζία και η Οσετία στη Γεωργία θεωρούμε ότι είναι ορθός ο χαρακτηρισμός κατεχόμενα εδάφη πρόκειται άλλωστε για ανακοίνωση προς τη Γεωργία πρέπει να τροποποιηθεί η αρχιτεκτονική της ασφάλειας και να μην χρειάζεται πλέον η επιβολή βίας. Οι δικές μου τροπολογίες κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον ε, τομέα της δικαιοσύνης. Επιταχύνθηκαν οι δίκες, αλλά χρειάζεται ακόμα να γίνει βελτίωση, κυρίως αν θέλουμε να μιλούμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό που θεωρώ ότι είναι προβληματικό και όπου πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή απέναντι στην μικρή εγκληματικότητα. Πάντως κρατούνται πολλοί στις γεωργιανές φυλακές. Οι συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές αυτές είναι εντελώς ακατάλληλες, ή δε κρατούμενοι κρατούνται εκεί για υπερβολικά μακρά διαστήματα σε σχέση με τις, με τις άδικες πράξεις που έχουν διαπράξει. Επίσης υπάρχουν περιορισμοί στις επαγγελματικές δραστηριότητες ορισμένων. Ασκούνται πιέσεις Γίνονται κάποιες πρόοδοι στην ε, οικοδόμηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά πρέπει να παρακινήσουμε τη Γεωργία να δείξει να επιταχύνει το βήμα και στον τομέα της δικαιοσύνης. Έχουμε και τον εργατικό νόμο, δεν είναι σαφές τι κάνει η γεωργιανή κυβέρνηση. Διευκολύνονται οι απολύσει. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της αποφυγής των διακρίσεων και σε ό,τι αφορά βέβαια τα συνδικαλιστικά δικαιώματα πρέπει κάτι να γίνει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Γεωργία πρέπει να γίνει σεβαστή η ελευθερία των μέσων, πρέπει να έχουν την ελευθερία να ενημερώνουν, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πιέσεις. Έχει ψηφίσει σημαντικά νομοθετήματα η Γεωργία στον τομέα. Αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη όμως για πλήρη ελευθεροτυπία όταν ακόμη διεξάγονται δίκη σε βάρος δημοσιογράφων. Ακόμα δεν έχουν βέβαια εκδοθεί αποφάσεις, αλλά έχουν υπάρξει και φόνοι δημοσιογράφων. Θα συζητήσω πάντω και με, και με τον εισηγητή και του άλλου και οδησηγητές για να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε. Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση του. Συνεργαστήκαμε μέχρι την πρώτη παρουσίαση της έκθεσης. Ε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, Σίγουρα πρόκειται για μια νέα ισορροπημένη και κατά τη γνώμη μου ορθή προσέγγιση που υιοθετεί ο εισηγητής γιατί η Γεωργία έχει τις ε, καλύτερες επιδόσεις ε, από την ανατολική εταιρική σχέση. Βεβαίως ε, υπάρχουν διάφορα ζητήματα υποσυζήτηση δηλαδή για ολοκλήρωση ή για συνεργασία. Τι επιθυμούμε ακριβώς, πώς επιθυμούμε να μετεξελιχθεί η σχέση μας με τη χώρα εγώ θα έλεγα ότι το πιο ρεαλιστικό θα ήταν να μιλήσουμε για ολοκλήρωση. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Λίζεκ που ε, δεχτήκατε την ε, πρότασή μας για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών αυτών, δηλαδή την παράγραφο 1. Σίγουρα, εάν θέλουμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, αν θέλουμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα θα πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία με την ε, Ρωσία ε, ούτως ώστε να ασκήσουμε πίεση για την ε, περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων. Επίσης, θα θέλαμε να εντατικοποιήσουμε την συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και τη Γεωργία. Η τροπολογία μας 15 δηλαδή ενδέχεται να ε, καταλήξουμε και συμβαστικές τροπολογίες. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα, διότι είναι παρεμφερείς ε, πολλές ε, από τις τροπολογίες. Καλωσορίζω την 539 και 45 σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις για την ενευτική διαδικασία, για το διάλογο τώρα με την αντιπολίτευση. Είναι σημαντικό ε, για τη χώρα να προαγάγει έναν ουσιαστικό πλουραλισμό και να ενισχύσει το διάλογο με την αντιπολίτευση. Τώρα, σχετικά με την ανάγκη ενός ανεξάρτητου δικαστικού ε, συστήματος, ε, φυσικά συμφωνούμε πάντως. Υποστηρίζουμε το σύνολο της έκθεσης και το όραμα που, του κ. Λίζεκ που απηχεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Λούνετσεκ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον εισηγητή. Η έκθεση αυτή ε, είναι μια καλή βάση και ευχαριστούμε που είστε πρόθυμος να συζητήσετε μαζί μας. Ούτως ή δεν υπάρχουν και τόσο πολλές τροπολογίες. Νομίζω ότι εύκολα θα καταλήξουμε συμφωνία για τις περισσότερες από αυτές. Ε, συγκεκριμένα αυτό που μου αρέσει είναι ε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της ολοκλήρωσης Ουκρανίας, δηλαδή της προσχώρησης Ουκρανίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προδικάζεται το τέλος. Δεν, ήταν, δεν είναι και το αντικείμενο της έκθεσης. Στην ε, τελευταία σύνοδο κορυφής εκεί μιλήσαμε για πολιτική σύνδεση ε, και οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρούμε αυτή τη φρασιολογία. Ζητώ συγγνώμη, κάντε φασαρία, λέει Μιλήτρια. Ε, συμφωνώ με αυτούς που διαχωρίζουν τη θέση τους για την Νότια Οσετία και την Απχαζία ότι θεωρούν ότι είναι κατεχόμενα εδάφη. Πιστεύω ε, ότι η στάση της χώρας είναι σαφής. Καλό θα ήταν ε, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή ε, πολιτικά και στρατιωτικά. έχει υποστηρίξει η Ρωσία τις τοπικές αρχές και έχουν παραβιάσει την κεχηρία. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τις προσωρινές διοικητικές αρχές, απλώς να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Γι' αυτό και υπέβαλα όλες αυτές τις τροπολογίες. Ε, κατόπιν οι σε για την ενότια ως αιτία Εκεί ονομάζεται νότια περιοχή Τσίχαν βάλει, δεν ξέρω και αν το προφέρω σωστά. Ε, συμφωνώ με αυτές τις τροπολογίες πάντως και θα λάβετε και μία δική μου σχετική. Τώρα τα θέματα ε, που σχολίασε η Τάνια Φαγιών με βρίσκουν σύμφωνοι και με, τα συμπεριλαμβάνω και σε κάποιες ε, τροπολογίες μου. Όντως, ε, διαπιστώνω και εγώ πρόοδο στο θέμα της κατάργησης κριτικής μεταχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μεταρρύθμισης του δικαστικού σώματος κτλ. Ε, το δέχομαι, αλλά αλλά υπάρχουν ω προς την υλοποίηση των μέτρων και ζητήματα που οφείλουμε να εξετάσουμε διεξοδικότερα. Ξέρω ότι η γεωργιανή κυβέρνηση δυσκολεύεται να το δεχτεί αυτό, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι ως Ευρωπαίοι πολίτες το οφείλουμε στους πολίτες της γεωργίας να με διαφάνει δηλαδή να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα. Η τροπολογία 38 της Τάνια Φαγιών, παραδείγματος χάρη, μιλάει για πρόσφατες υποθέσεις ε, ε, δικηγόρων που δέχτηκαν επίθεση και κακοποιήθηκαν από αστυνομικέ δυνάμεις. Συγγνώμη, αλλά ως Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουμε να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και να ξεκαθαρίσουμε στις γεωργιανές αρχές ότι ε, κάντε κάτι, ερευνήστε τις υπόθεσεις και με σαφή να αναδείξετε ότι το αστυνομικό σας σύστημα δεν παρεμβαίνει στην διερεύνηση δικαστικών υποθέσεων. Τώρα, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εκεί ε, πολλά υπολείπονται ως προς και για την υποστήριξη της δράσης τη κοινωνίας των πολιτών. Ε, είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω θα καταλήξουμε σύμφωνοι για αυτό το θέμα. Τώρα, τροπολογία 32, δική μου τροπολογία. Για ιστορικούς λόγους, για όλα αυτά που έχουν συμβεί, πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρουμε πως ε, λυπούμαστε που έγινε μία πρόταση, μία επίθεση πριν το 2008, πριν ε, να εισβάλλει στρατιωτικά η Ρωσία και ο Σακασβίλη την απέριψε. Ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό, δηλαδή τι έγινε πριν τη ρωσική εισβολή και κατόπιν κατοχή. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και Προσβλέπω με ανυπομονησία στις ε, λατικές συζητήσεις μας για τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε κύριο Σκόρνιτσεκ. Ευχαριστώ. Ακούγοντας ορισμένες συναδέλφους, ευνηδιάζομαι γιατί μιλούν για κατεχόμενα εδάφη. Ενώ από την άλλη μεριά διαρριγνούν τα μάτια τους υπέρ του ελεύθερου Κωσόβου. Αν εξετάσουν τις τροπολογίες, την τροπολογία παριθμών ένα, για παράδειγμα, του κ. Λαντσμπέργκης λέει ότι η Γεωργία είναι ευρωπαϊκή χώρα που οικοδομεί επιτυχώς τη δημοκρατία. Ο ίδιος, ωστόσο, Λαντσμπέργκης λέει σε άλλη τροπολογία ότι ορισμένα εδάφη αποτελούν θυμά της γεωργίας. Αυτό αποτελεί ωστόσο αντίφαση. Μπορώ να πω και ότι το Ισλάμ και ο χριστιανισμός έχουν κοινέ ρίζες. Αλλά δεν μπορώ να βγω και να πω ότι το Τιδό είναι χριστιανική χώρα. Και ότι θα πρέπει να προσαρτηθούν σε αυτήν οι Ισλαμικές περιοχές. Για τη Γεωργία βλέπω το πρόβλημα ότι υπάρχουν, λειτουργούν κανόνες σε διαφορετικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία και για την εφαρμογή των κανόνων που είναι η συνήθι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι κανόνες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, για παράδειγμα, εφαρμόζονται σωστά. Λυσμονούμε ότι η Γεωργία έχει και γείτονες και δεν μιλούμε καθόλου, για παράδειγμα, για την σχέση της Γεωργίας και της Τουρκίας, της Γεωργίας και της Αρμενίας. Δεν μιλούμε καθόλου στο ψήφισμα αυτό. Αλλά αυτά είναι σημαντικά. Όταν θέλουμε να διαπραγματευτούμε με κάποιον και θέλουμε να προσεγγίσει η χώρα αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξετάσουμε και τις γειτονικέ της σχέσεις και αυτές να είναι κρυσταλλίνες διαβιές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ειρηνικέ σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες. Βλέπω ότι υπάρχουν 30 τροπολογίες που αναφέρονται στη σχέση με τη Ρωσία. Εγώ δεν θα σχολιάσω καθόλου εάν πρόκειται για περιοχές οι οποίες ανήκουν στη Γεωργία ή όχι. Αλλά η Γεωργία είχε ζητήσει τη βοήθεια της Ρωσίας όταν βρίσκεται σε σύγκρουση με την Τουρκία. Ε, τότε να πούμε ότι η Γεωργία είναι μέρος της Τουρκίας και άρα γιατί συζητούμε. Είναι απαραίτητο να εφαρμόζουμε ίδια κριτήρια για τις χώρες που βρίσκονται στα πλαίσια της προσανατολάς γειτονίας. Και για τη Γεωργία θα πρέπει να εφαρμόζουμε πάντοτε τα αυτά μέτρα και σταθμά. Και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα δημοκρατικά στοιχεία που διαλαμβάνονται και σε άλλες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα εκμεταλλευτώ και εγώ αυτή την ευκαιρία για να αναφερθώ στα συμβάντα της Γεωργίας. Κάποια στοιχεία εντοπίστηκαν ήδη από τον εισηγητή, αλλά θα ήθελα να τα σκεφτούμε και με ένα κριτικό πνεύμα. Το θέμα είναι να δούμε σε μια πρώτη φάση πώς ε, τοποθετήθηκε το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε πώς αποτιμά την κατάσταση το πολιτικό σύστημα. Αν δούμε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην ε, Γεωργία, τις οικονομικές εξελίξεις, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά θα είναι καθοριστική σημασία για να δούμε την απόκριση που μπορούμε να δώσουμε έπειτα. Κατά πόσον, ε, πρέπει να δούμε κατά πόσον η Γεωργία είναι έτοιμη να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Οδό. Μιλώντα με πολιτικού ευθύνοντε από την Γεωργία και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω ότι αυτή η διασύνη προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέγγιση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διαρκής και αυξανόμενης έντασης αλλά εδώ φαίνεται ότι οι προθέσεις των Γεωργιανών για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιούνται και στην πράξη. Κυρία Όγιολαν, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με αυτών των συναδέλφων που συνεχάρισαν τον εισηγητή. Και να προσθέσω κάτι στα σχόλια που ακούσαμε. Για το θέμα αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι, πώς θα βαρύνει η έκθεσή μας αυτή και θα επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα στη Γεωργία. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε τις πολιτικές παρατάξεις που μπορεί να διαφωνούν, να σκεφτούν την προοπτική της Ευρώπης. Διότι υπάρχει και η προοπτική της Συμφωνίας Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών και θα πρέπει η Γεωργία να καταλάβει ότι το χρειάζεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται και άλλο εμπόριο και ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθούν οι πολιτικέ παρατάξει στη Γεωργία να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους να προσεγγίσουν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους. Η επόμενη παρατήρησή μου έχει να κάνει με το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Και εδώ θα πρέπει να δούμε την προοπτική που χαράσει η έκθεση αυτή. Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά το κείμενο, νομίζω ότι θα αντιληφθεί ότι η έκθεση συνολικά μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Γεωργίας. Δηλαδή, πέραν των σύνορων της χώρας, ενθαρρύνοντας και τις γείτονες να ακολουθήσουν το επιτυχές παράδειγμα της Γεωργίας, οι πλησιέστεροι γείτονες όπως η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά και τα κατεχόμενα εδάφη και το ρόλο που διαδραματίζει η Ρωσία στην Γεωργία. Εδώ θα ήμουν ακόμη πιο αυστηρή από τη έκθεση. Δηλαδή δεν θα έκανα απίθυνα απλώ έκκληση στην Ρωσική Ομοσπονδία να ακολουθήσει και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις ώστε να πάψει την κατοχή της Νότιας Οσετίας και της Απχαζίας. Θα το εξέφραζα ως απέτηση από την ε, Ρωσική Ομοσπονδία να αναλάβει τι διεθνεί τη υποχρεώσει. Ευχαριστούμε, κύριο Λίσεκ. Για να κλείσουμε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για να μην σα καθυστερήσω. Σα ευχαριστώ όλου για τι παρεμβάσει. σα. Θα διαπραγματευτούμε και πάλι βέβαια τις τροπολογίες, όπως είπα, είμαι πεπισμένος μετά και από την συζήτηση που μόλις διεξήχθη, ότι θα βρούμε συμβαστικές λύσεις. Ο κ. Κόβαλ έθεσε μια ερώτηση που νομίζω ότι δεν είμαι σε θέση να την απαντήσω γιατί είμαι εισηγητής. Αλλά η δεύτερη, θέση, η δεύτερη ερώτηση που έθεσε είναι περισσότερο ερώτηση προς, που θα έπρεπε απευθυνθεί στην Γεωργιανή ηγεσία. Ο κύριος Κόβαλ γνωρίζει τους αρμόδιους πολιτικούς και νομίζω σε αυτούς θα έπρεπε να απευθυνθεί. Συμφωνώ ωστόσο με αυτό που λέει ότι πολλά κινούνται με υπερβολική βραδίτητα στην Γεωργία και θεωρώ ότι πολλά θέματα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Και γι' αυτό στην έκθεσή μου αναφέρω ότι χρειαζόμαστε κοινή θέση όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και πολλές ερωτήσεις βέβαια να απαντηθούν σύντομα. Σε ό,τι αφορά την αποφασιστικότητα των Γεωργιανών, κατά πόσον είναι δηλαδή σε θέση να αναμείνουν ακόμα και πώς θα, πόσο θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους τα θεσμικά όργανα. Αυτή την ερώτηση θα μπορέσουμε να την κάνουμε στις 19 Οκτωβρίου όταν θα προσέλθει εδώ ο πρόεδρος της Γεωργιανής Βουλής. Μπορούμε τότε να του κάνουμε απευθεία την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την αντιπολίτευση, η και με αυτό που εσείς αποκαλείτε υπερβολικά αργή εξέλιξη στην δημοκρατική οικοδόμηση, εν μέρει συμφωνώ μαζί σας. Ασφαλώς υπάρχουν ορισμένα θέματα που ίσως να μην ε, αφορούν τόσο πολύ τις πιο πρόσφατες εκλογές, αλλά τις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχε γίνει τότε και αποστολή παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχα την τιμή να συμμετέχω, η κυρία Νικολάη επίσης. Στις τελευταίες εκλογές δεν φάνηκε να υπάρχει λόγο να διατυπωθούν σημαντικές μομφέ. Λόγω τη εισηγήσεώ μου πήγα τρει φορές στη Γεωργία, συναντήθηκα με όλους τους πολιτικού σχηματισμού. και με αυτούς που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο αλλά και με την εξοκοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Μίλησα και με τις μειονότητες, με εκπροσώπους γερμανικών, αγγλικών και γαλλικών ιδρυμάτων και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα, ότι η Γεωργία βαδίζει στην σωστή κατεύθυνση. Είναι δημοκρατία. Το κόμμα του Προέδρου Σακασβίλη κερδίζει τις εκλογές και έχει και δύο τρίτα των ψήφων, των εδρών μάλλον στη Βουλή. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει στην βάση βίας και νοθείας. Αλλά από, οφείλεται στο γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι διαρεμένη και αδύναμη. Το ίδιο για το αξίωμα του Δημάρχου της Τυφλίδος, όπου υπήρχαν 10 υποψήφοι και αυτοί οι δέκα υποψήφοι μισούσαν οι μεν τους δε. Ήταν αδύνατο να συνεργαστούν μαζί τους, μεταξύ τους. Και αυτό βέβαια ωφελεί το κόσμο του Σακασφίλη και τους υποψηφίους του. Πρέπει άρα να είμαστε συνεπείς, να υποστηρίξουμε τη γεωργία πολιτικά, οικονομικά, χρηματοδοτικά και αυτό προσπαθώ να εκφράσω και με τη σύστασή μου. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην περαιτέρω εξέλιξη της δημοκρατίας στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Πριν ξεκινήσουμε και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λεγκούτκο, να σας θυμίσω τρία πράγματα. Πρώτον, το πρωί, σε αυτή την αίθουσα, είχαμε έναν υπουργό Εξωτερικών και συζητήσαμε μαζί του. Έπειτα, σήμερα, κατά τη συζήτηση αυτή, ανακοινώθηκε επισήμω ότι η Γιώτη Μοσέμκο καταδικάστηκε σε επταετή κάθριξη και το τρίτο στοιχείο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η απόφαση της ΙΝΤΑ ήταν να αναβληθεί η ψηφοφορία τους ε, για την ε, σχετική γνωμοδότηση. Τα τρία αυτά στοιχεία θέλουν να τα έχετε υπόψη πριν πρώτο ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε Λεγκούτκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω όλους τους και εισηγητές και συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. 140 περίπου τροπολογίες και μας διευκόλυναν στη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης. Ο διάλογος ήταν διαρκής και επικοδομητικός. Υπάρχουν κάποια σημεία βέβαια που απομένουν να συζητηθούν. Θα το συζητήσουμε στο προσοχές μέλλον, όμως θεωρώ ότι φτάσαμε σε κάποιες καλές συμμεμπαστικές λύσεις. Η κατάσταση στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή ε, εξελίσσεται και μεταβάλλεται διαρκώς με πολύ δυναμικό τρόπο. Προσφάτες, ε, εξελίξεις υπάρχουν διαρκώς μάλλον, ακόμη και προσ, προσφάτως και κάποιες οπισθοχωρήσεις δυστυχώς. Ξέρουμε όμω πόσο σημαντική είναι η Ουκρανία στι σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο μα ενδιαφέρει να διατηρούμε θερμέ σχέσει με τη χώρα αυτή. Οι διαφωνίε μα αφορούν τα μέσα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να μετέλθουμε για να πετύχουμε κοινού στόχου. Αλλά και ω προ του στόχου διαφωνούμε μεταξύ μα. Οι στόχοι λοιπόν είναι οι καλές σχέσεις η οικοδόμηση ενός δημοκρατικού σταθερού κράτους στην Ουκρανία που να σέβεται τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, που να έχει ένα πλήρες δικαστικό σύστημα, να προστατεύει τις μειονότητες. Βασικές προδιαγραφές αυτές. Οποιασδήποτε σύγχρονης συνταγματικής δημοκρατίας. Πριν από την συμφωνία σύνδεσης, θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός διάβλος για την ε, ε, ολοκλήρωση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας και βεβαίως για τη μελλοντική προσχώρηση ενδεχομένω της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Για τους περισσότερους Ουκρανούς, νομίζω για την πλειονότητά τους, η προοπτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να μοιάζει με φως στην άκρη του τούνελ. Γι' αυτό συζητήσαμε διαμακρών την πρόπτικη αυτή, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συστηματικές και εντατικότατε μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει και αυτή τη στιγμή ε, εξάγονται σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει όμως αυτή η προσπάθεια να εξακολουθήσει. Το πλαίσιο το παρέχει η σχετική συμφωνία για τον εξυγχρονισμό του Ουκρανικού κράτους καθώς και ο σχετικός οδικός χάρτης. Βεβαίως, πέραν όλων αυτών των στοιχείων, να σταθώ και εγώ στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Προέδρου ε, για το τι συνέβη σήμερα. Δεν ήταν καλή μέρα για μας και τους φίλους της Ουκρανίας. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να συλλογιστούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα πρέπει να κάνουμε σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Θα συναντήσω αύριο τους συνεισηγητές και θα τους προτείνω την αναβολή της πληροφορία. Και αυτό προκειμένου να, διατηρήσουμε, να τηρήσουμε μάλλον μια συνετότερη και ορθολογικότερη στάση προκειμένου για το επόμενο βήμα μας. Ευχαριστώ. Επειδή δεν θα είστε για πολλή ώρα μαζί μας, θα σας δώσω το λόγο και κατόπιν στον επόμενο συνάδελφο. Ναι, ο εισηγητής με κάλυψε Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τώρα ασφαλείς προβλέψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Υπονομεύονται αυτή τη στιγμή όλες μας οι συμβαστικές λύσεις. Οπότε θα στηρίξω την πρόταση του εισηγητή για αναβολή. Προέδρε, ευχαριστούμε. Κύριο Κόβατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Λεγκούτκο για την πρότασή του. Πράγματι και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να επαναθεωρήσουμε τις συμβαστικές μας λύσεις, ιδίως την 2, 4 και την 5, υπό το φω των προσφατότερων πληροφοριών. Κατά τα άλλα, σημερινέ ειδήσει δεν αλλάζουν την πραγματικότητα τη Ουκρανία. Η Ουκρανία χρειάζεται την Ευρώπη και το αντίστροφο. Όμω δεν πρέπει να διαπράξουμε το σφάλμα. Ένα, βρα... Ένα σφάλμα εδώ, ξεχνώντα ότι η Ουκρανία που χρειαζόμαστε πρέπει να είναι δημοκρατική, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με δικαστικό σύστημα, με δημοκρατικό καθεστώ. όχι να οδεύει προς την απολυταρχία. Ε, η δική μου επιθυμία είναι να γίνει εξόπιστο εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία και ελπίζω ότι θα εμβαθύνουμε τι σχέσει μα ώστε να υπάρχει αμοιβαίο όφελο και για του Ουκρανού πολίτε και για του Ευρωπαίου. Ε, πολίτε ε, τη Ουκρανία που όμω θα ζουν σε ένα πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα θεσμικά όργανα να εργαστούν προκειμένου να, να έρθει πίσω στην δημοκρατική οδό αυτή η χώρα. Σήμερα ήταν πολύ παράξενο, ειδικά για μένα, που την ίδια μέρα ένας εκπρόσωπος μιας συγκεκριμένη χώρας ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας για να μας πείσει ότι ακολουθούν όλους τους δημοκρατικούς κανόνες, ενώ ταυτόχρονα έφτανε η γνωστή είδηση στα αυτιά μας. Ήταν πολύ ατυχές αυτό. Το αντίθετο ελπίζαμε. Ελπίζαμε να έχουμε πολιτικές ενδείξεις από την Ουκρανία ότι αυτό δεν θα συμβεί. Αυτό που επιθυμούσαμε να μην συμβεί. Όμω ε, προσδοκούμε και εμεί τη συνάντηση με του σκεώδει εισηγητέ και θα σα ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα. Πρώτα. ευχαριστούμε. Δύο τελευταίοι εισηγητές. ο κ. Σούλτ Με τη σειρά μου θα ευχαριστήσω τον κύριο Λεγκούτκο, ο οποίος δέχθηκε να επεξεργαστεί τις περισσότερες από τις προτάσεις μας για δημοκρατία κλπ. Κύριε Λεγκούτκο, είπατε ότι θα πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας περισσότερο χρόνο. Και εγώ είμαι υπέρ της αναβολής της εκθέσεως. Αυτό αναφέρεται όμως και στον Συμβασμό 5, ότι θα πρέπει να διαθώσουμε περισσότερο χρόνο. Και οι διαπραγματεύσει δεν πρέπει να τελούν υπό πολιτική πίεση. Δεν ε, υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε ε, κάποια προθεσμία μέχρι τέλους του έτους, για παράδειγμα, για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις. Σήμερα είδαμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση που μας διδάσκει ακριβώ το αντίθετο. Διότι σήμερα πραγματικά ήταν προσβολή. Ούτε πιστεύω ότι ήταν σύμπτωση ότι σήμερα προσήρθε ο Υπουργό των Εξωτερικών και αυτή η είδηση τον πέτυχε, τον έπληξε πισόπλατα. Στην ουσία αυτό που ήρθε και μας είπε είναι ότι μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Θα διώξουμε την αντιπολίτευση, θα την κατατροπώσουμε την αντιπολίτευση και υπό τις συνθήκες αυτές νομίζω ότι όντως χρειάζεται να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στους εαυτούς μας. Ευχαριστώ Κόβατσεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Κόλιτσεκ. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Σούλτς. Ίσως στη δική του χώρα να είναι δυνατόν να επηρεαστεί ένα δικαστήριο από πολιτικές πιέσεις πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ουκρανία. Σίγουρα θα γνωρίζετε και πολύ καλά αυτά που πρότεινε ο Ουκρανός Πρόεδρος ότι για οικονομικά εγκλήματα κανείς δεν θα εγκλειστεί στις φυλακές. Και αυτή η απόφαση λήφθηκε και στο Κοινοβούλιο. Αυτό όμως δεν το είπε ο υπουργό, τουλάχιστον όχι έτσι επιλέξει. Ολόκληρη αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι όλα έχουν α, εδώ προπαρασκευαστεί καλώς, βλέπω να λείπουν κάποια τεχνικά θέματα, μιλούμε για τον αγωγό αερίου καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια για τα οποία είχαμε μιλήσει και σε ένα ψήφισμα και είχαμε πει τότε ότι καλό θα ήταν να συνεργαστεί η Ουκρανία και με τις γειτονικές χώρες και βεβαίως αυτό θα είναι επιθυμητό και είναι προκειμένο. Βασικά πάντως αυτό που ενδιαφέρει είναι η μεταφορία του φυσικού αερίου και εδώ δεν περιλαμβάνεται. Στις 142 τροπολογίες αυτές ασφαλώς πρέπει να κρυθούν, να εξεταστούν προσεκτικά και με όλο τον απαραίτητο χρόνο. Ας μην λησμονούμε όμως ότι διαπραγματευόμαστε ταυτόχρονα με όλους τους γείτονες, με όλες τις γείτονες χώρες. Και η Ουκρανία πραγματικά βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες θέσεις σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Συνδέσεως. Ο κύριος και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις ορισμένων συναδέλφων. Οφείλω να ομολογήσω ότι τις τελευταίες εβδομάδες ασχολήθηκα πολύ με το θέμα αυτό της νομιμότητας των δικών και την πρόοδο της Συμφωνίας Συνδέσεως. Και πίστεψα επίσης ότι από ουκρανικής πλευράς θα αντιλαμβάνονταν την αξία αυτών των συσχετισμών. Σήμερα ωστόσο το δίδαγμα ήταν διαφορετικό. Τα πράγματα δεν έγιναν ευκολότερα για μένα σήμερα. Και με καθιστά αβέβαιο. Δηλαδή η θέση μου πλέον δεν είναι τόσο η θέση την οποία είχα δεν είναι πλέον τόσο ε, σίγουρη, δεν είμαι τόσο σίγουρος για αυτήν. Διότι βεβαίως η Ουκρανία είναι σημαντικό στρατηγικός εταίρος. και είναι σταυροδρόμοι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Υπάρχει η δυνατότητα ίσως την επόμενη Τρίτη στην δεύτερη στην δεύτερη ε, ανάγνωση του νομοσχεδίου στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο να γίνει κάτι. Επίσης η επίσκεψη Γιαννουκόβιτς που μάλλον τώρα δεν θα γίνει γιατί ο Μπαρόσο βρίσκεται εδώ. Ας μην βιαστούμε λοιπόν. Είχα προτείνει επίσης, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια και να κάνει μια δήλωση η κυρία Κάθη Άστον για, το, για την υπόθεση Τιμοσένκο και α ορίσει κάθε πολιτική ομάδα έναν αγορητή. Α μην κάνουμε ψήφισμα ακόμα, ίσω να το κάνουμε στο Στρασβούργο τον Νοέμβριο. Αλλά α συζητήσουμε το θέμα αυτό μεταξύ μα. Α δώσουμε ξεκάθαρα μηνύματα που νομίζω ήδη δόθηκαν ξεκάθαρα σήμερα στον Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι κατενόησε την σημασία της έννοιας κράτος δικαίου. Για να μιλήσουμε για κράτος δικαίου θα πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνουν τι εννοούμε. Ότι όλα δεν έχουν ολοκληρωθεί βεβαίως τα γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση ότι κάνουν πορεία προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και στη Μολδαβία και στη Γεωργία τα πράγματα δεν έχουν καταλήξει ακόμα, αλλά έχω την εντύπωση τουλάχιστον ότι πηγαίνουν προς την κατεύθυνση παρόλε τι κριτικέ. Και οι Ουκρανοί που ήταν σε καλό δρόμο, ειδικά σε αυτό το θέμα τώρα της, των δημοκρατικών αξιών του κράτου δικαίου, δεν τα πάνε καλά. Και αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί κανεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπολογίζουμε, δεν θέλετε να, να ξεπουλήσετε την οικονομία σας στη Ρωσία, αυτό ναι, αλλά τότε πουλούμε εμείς την ψυχή μας. Γι' αυτό και πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους, να προσφέρουμε και τρόπους και στην Ουκρανία να μπορέσει η ίδια να ξεφύγει από την κατάσταση αυτή. Οι ίδιοι πρέπει να βρουν τους τρόπους. Αν όμως δοθούν μηνύματα εδώ από το ευρύ πολιτικό φάσμα, όπως αυτά που ακούστηκαν σήμερα, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε κάποιες εξελίξεις. Και αν συμφωνεί ο συνάδελφος εισηγητής, μπορούμε ίσως να το περιλάβουμε και σε κάποιες τροπολογίε αργότερα. Να ξανασκεφτούμε αν ίσως ξανανοίξουμε προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών. Για να μπορέσουν και οι συνάδελφοί μας της ΙΝΤΑ με τον τρόπο αυτό να ε, ολοκληρώσουν την γνωμοδότησή τους κάτι που δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν. Αν συνεχίσουμε με business as usual, νομίζω δεν τιμούμε το θέμα. ώστε να περιλάβουμε και την προστασία της αντιπολίτευσης. Ευχαριστούμε κύριο Γιόλαντ. Ευχαριστώ. Ε, η αναβολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία δεν συνιστά κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί συνάδελφοι σήμερα έχουν σοκαριστεί, ε, είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και ίσως είναι λογικό να αποφασίσουμε μια σύντομη αναβολή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Γνωρίζοντα όμω αυτή τη χώρα με όλη την περίπτωση κατάσταση που εκεί επικρατεί, είμαι απολύτω πεπισμένη ότι αυτό που συνέβη ε, σήμερα το πρωί δεν είναι τυχαίο, δεν πρόκειται για σύμπτωση. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάποιοι στη Μόσχα χαίρονται για τα όσα συνέβησαν σήμερα. Τις ε, περασμένες εβδομάδες συναντήθηκαν με διάφορους εκπροσώπους στο Κοινοβουλίο της Ουκρανίας ε, στο Στρασβούργο ε, και κάποιοι ήταν στη μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην πλευρά του συνασπισμού, δηλαδή του κυβερνητικού συνασπισμού. Πέρσι συναντήθηκα με πολιτευόμενους συνάδελφοι από τους φιλελευθέρους ήρθαν σε επαφές ανεξαρτήτως πολιτικές θέσεις είτε συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό είτε όχι ε, και συζητήσαμε και για την υπόθεση Τιμοσέγκο και ε, ε, φυσικά ε, παρόδο πρέπει να ληφθεί απόφαση από ανεξάρτητο διεθνές δικαστήριο. Ε, Πάντω για τι συμφωνίε σύνδεση θα πρέπει να διατηρηθεί και γιατί και τα δύο μέρη επιθυμούν την προσχώρηση της χώρας Δεν θέλουν να πέσουν και πάλι στον έλεγχο της Μόσχας και ξέρετε πόσο μεγάλη πίεση ασκεί η Ρωσία, μετέρχεται διαφόρων μέσων για να επιτύχει το στόχο της ε, με καλούς αλλά και κακούς τρόπους ε, προσπαθεί ε, να σπρώξει την Ουκρανία σε τελωνιακή ένωση με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν. Αυτό είναι το βασικό θέμα και αν εμείς δεν τον αντιλαμβανόμαστε από πολιτικής πλευρά ζητώ συγγνώμη αλλά θα πάρουμε λάθος απόφαση. Decisions uh, and... Uh, ε, τις ε, δηλώσεις που ακούσαμε σήμερα και τα όσα συνέβησαν σήμερα, ελπίζουμε ότι τελικά θα φανούμε ρεαλιστές εδώ στην Ευρώπη και θα κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ανατολική γειτονική χώρα. Ο κύριος Πάσκου την εντύπωση ότι κάπου είδα στον τύπο ότι δεν ευχαριστήθηκε, δυσαρεστήθηκε μάλλον η Ρωσία από την απόφαση του Κιέβου. Τέλος πάντων. Ο κύριος Ζαλεύσκη, ε, πρόεδρε, ε, είμαι εισηγητής ε, της ε, ΙΝΤΑ για την καθολική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, τη σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και με αυτή την ιδιότητα παίρνω το λόγο θα ε, μπορούσατε να εξετάσετε τον ενδεχόμενο αναβολή στις ψηφοφορίες στην Επιτροπή Αφέτη για το ψήφισμα σας το ζητήσαμε διότι θέλαμε να ψηφίσουμε στη δική μας Επιτροπή σήμερα. Άρα είναι σημαντικό να ε, συντονίσουμε τα χρονοδιαγράμματα εργασίων των δύο επιτροπών. Νομίζω ότι όλοι σοκαρίστηκαν από την καταδικαστική αυτή απόφαση ε, είναι η ανώτατη μέγιστη ποινή βάση του ε, Ουκρανικού ποινικού κώδικα που προβλέπεται για αυτή την αξιόπινη πράξη και σήμερα ε, είναι σημαντικό όλοι όσοι εδώ στο Κοινοβούλιο ε, επιθυμούν ε, την προσέγγιση της Ουκρανίας και την προσχώρηση της στην Ένωση. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι σημαντικό να ε, στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις Ουκρανικές αρχές ότι δεν θα δεχτούμε την παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων. Επίσης να περάσουμε το μήνυμα ότι έχουμε βαρεθεί πια, έχουμε βαρεθεί με αυτές τις αποφάσεις των Ουκρανικών αρχών και δεν σας μιλώ τώρα για την δικαστική απόφαση γιατί δεν θέλω να ε, μπω σε αυτή ε, τη συζήτηση. Πρόκειται για τη σχέση ανάμεσα στα δικαστήρια και τις αρχές. Ε, τέλος πάντων, την περασμένη εβδομάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου έγινε συζήτηση για την ποινικοποίηση κάποιων άρθρων του κώδικα, μεταξύ των οποίων και αυτό ε, το οποίο επικαλέστηκε η δικαστική αρχή για να εκδώσει την απόφαση κατά της κυρίας Τιμοσέγκου και δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι να πούμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνία. Οι πολίτες ε, της Ουκρανίας και αυτή η συμφωνία σύνδεσης, αυτή η σφαιρική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, αυτούς θα ωφελήσει τους πολίτες της Ουκρανίας. Και έχουμε βαρεθεί πια που ε, οι αρχές ε, Ε, θυσιάζουν το συμφέρον ε, των ε, πολιτών στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα σας ευχαριστούμε κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ χωρίς καμία αμφιβολία. Όλους θα πρέπει να μας απασχολεί η έννοια του κράτους δικαίου. Θα Χαιρόμουν πάρα πολύ αν αυτό συνιστούσε προτεραιότητα και στις ε, σχέσεις ε, ε, ανάμεσα στα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι στη Ρουμανία είχαμε αντίστοιχα προβλήματα με την αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί ένα τέτοιο νομικό ζήτημα μας με εμποδίζει από το να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία σύνδεση, να εξετάσουμε τι ε, μελλοντικέ μα σχέσει με την Ουκρανία. Μα είναι προ όφελο και των δύο μερών η συμφωνία. Η δίκη της ε, κυρίας ε, Τιμοσέγκου θα επιληθεί βάσει της Ουκρανικής... Ε, ε θα ολοκληρωθεί βάσει της ε, Ουκρανικής νομοθεσίας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία, διότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενη η δίκη. Ε, αν τώρα θέλουμε, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες, εντάξει, να βάλουμε την ψηφοφορία, αλλά αυτός θα ήταν ε, ο σωστός λόγος για αναβολή. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία λόγω συναισθηματικών ε, αντιδράσεων ε, ή λόγω των όσων συνέβησαν σήμερα στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπερασπιστεί κάποια συγκεκριμένα άτομα και στις σχέσεις μας με τις ανατολικές χώρες θα πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα τη συνολική μας σχέση με όλους τους πολίτες της Ουκρανίας και όχι με συγκεκριμένες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής. Η έκθεση θα πρέπει να ψηφιστεί, θα είναι υποφελή η Σύμφωνια Σύνδεσης και για τα δύο μέρη ε, και δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο ε, λόγω της δίκης να αναβληθεί η ψηφοφορία. Μάλιστα σας ευχαριστούμε ο κύριος ε, Κόβαλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια για τη συμφωνία με την Ουκρανία. Όλες οι πολιτικές απόψεις ακούστηκαν εδώ και το ίδιο και στην Ουκρανία. Όταν διρωτώ με τα, κατά πόσον θα προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ομαλά, ε, ακούσαμε πολλές ε, διαφορετικές ε, απόψεις και ακούσαμε και το σχόλιο για την υπόθεση του Μοσέγκο ε, Στη συνάντησή μας με τον Υπουργό το συζητήσαμε αυτό, όμω βλέπουμε την κατάληξη και υπόθεση. Λοιπόν, νομίζω οι διαπραγματεύσει δεν πρέπει να ολοκληρωθούν ακόμη. Έχουμε ω το τέλο του χρόνου, ε, χρειαζόμαστε χρόνο για να σκεφτούμε και έχουμε την πολιτική διορατικότητα για να σκεφτούμε πώ θα εξετάσουμε το θέμα εν ευθέτω χρόνο και τι προτάσει μπορεί να προκύψουν. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ συναισθηματικοί εδώ. Καθώς πρόβλημα με την Ουκρανία έχουμε, αλλά δεν είναι επιπροσωπικού, είναι πρόβλημα με όλο το σύστημα της χώρας. Βεβαίως και οργιζόμαστε με αυτά που γίνονται. Όμως όλους συμφέρει και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινωνία της Ουκρανίας τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Κατά την ε, Πορτοκαλιά Επανάσταση είδαμε ποια ήταν τα αποτελέσματα των προσπαθειών, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις της Ουκρανίας το μόνο που επιζητούν σήμερα είναι να ολοκληρωθούν οι διπραγματεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερως επιφυλακτικοί. Να μην είμαστε συναισθηματικοί στις αντιδράσεις μας. Προφανώς το πρωί Είχαμε τον Ουκρανό εκπρόσωπο μαζί μας. Τέτοιου είδους εξελίξεις χρειάζονται χρόνο για να αφομοιωθούν. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε από τώρα τι πέρα θέλουμε να έχουν αυτές οι διαπραγματεύσει αίσιο ή όχι. Εάν η Ουκρανία λοιπόν θέλει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, εντάξει, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Θα ήθελα λοιπόν να βεβαιωθώ ότι θα αποφύγουμε βεβαιασμένες αποφάσεις. Κύριε Λαντσμπέργκης, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη μόνο παρατήρηση. Εάν οι ανησυχίες και επιφυλάξεις μας κατά της δίκης Τιμοσένκο οδηγήσουν σε αναβολή της συμφωνίας ε, ε, συνδέσεως με την Ουκρανία και εγγραφή στις ελληνικές καλένδες, τότε πρόκειται για τιμωρία. Και αυτό είναι σε βάρος ολόκληρης Ουκρανίας και του λαού της. Σε παρόμοιες συγκρίσιμες περιπτώσεις αυτό δεν το λησμονήσαμε, το είχαμε στο μυαλό μας. Για 30 δευτερόλεπτα ο κύριος Μπροκ. δεν είμαι βέβαιος τι στάση να κρατήσουμε. Να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις business as usual. Εγώ θα το εξαρτούσα αυτό από τις εξελίξεις των επομένων ημερών. Και ούτε θα ήθελα να ηγεθεί εντύπωση στην Ουκρανική κυβέρνηση ότι εδώ δεν πρόκειται να γίνει απολύτω τίποτα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκύψει ξανά την υπόθεση του χρόνου όταν θα τεθεί το θέμα τη κύρωση τη συμφωνία. Θα ήθελα να μπορέσει η Ουκρανική κυβέρνηση να βρει μια λύση που να επιτρέψει να βγει ασπροπρόσωπη και αυτή και εμεί. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πάσκου. Αναφέραμε εδώ. Βασικά καταγράψαμε τις βασικές απόψεις. Μία είναι να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Η άλλη είναι ότι να παρατείνουμε την ημερομηνία, ε, την προθεσμία υποβολή ε, ε, τροπολογιών και να έχουμε και νέες τροπολογίες. Η τρίτη εναλλακτική είναι να μην γίνει αυτό. Ο κύριο Κόβελ για 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δώσουμε ένα ξεκάθαρο, μονοσήμαντο πολιτικό μήνυμα. Οι διαπραγματεύσει έχουν δική του εντολή. Υπάρχει μια διαδικασία. Είναι επομένω τεχνική περισσότερο υπόθεση. Προ τη κυρώσεω και κατά τη διάρκεια τη κυρώσεω μπορούμε να προβάλλουμε πολιτικά επιχειρήματα και να θέσουμε πολιτικά θέματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφέ αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λεγκούτκο. Oh, <clears throat> Ευχαριστώ κυρίες ε, και κύριοι για όλα τα σχόλια και την υποστήριξη που μου προσφέρετε. Πιστεύω ότι ε, τέθηκαν διάφορα ζητήματα στη συζήτησή μας. Ε, το βασικό είναι Ποια θα είναι η σύστασή μα τελικά. Ε, συστήνουμε την, ε, ε, το πάγωμα των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία σύνδεσης ή την σύναψη της συμφωνίας. Εγώ δεν, προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συστήσουμε το δεύτερο, τη σύναψη της συμφωνίας δηλαδή. Όμως υπό το φω των πρόσφατων εξελίξεων που ε, βρήκαμε ότι είναι ανησυχητικές, ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε για να είμαστε σίγουροι, για να μην υπάρξει καμία παρανόηση. Βεβαίω είναι ε, κατανοητές οι αντιδράσεις, θα με εξέπλητε το αντίθετο. Πρέπει να ε, πάρουμε μια συνέτη, ξεκάθαρη απόφαση με αυτά τα ομολογουμένως αποκλίνοντα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και να συστήσουμε ενδεχομένως τη σύναψή της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης ε, για να περάσουμε το αντιαμφισβήτητο μήνυμα προς τις Ουκρανικές αρχές ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε τέτοιες κινήσεις όπως αυτές που ζήσαμε σήμερα, που βιώσαμε σήμερα. Συμφωνώ με ε, ε τα περισσότερα από αυτά που είπατε. Βέβαια υπήρχαν και αντιφάσεις ε, προφανέστατα. Όλοι πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από αυτά που συνέβησαν, αλλά το σημαντικό είναι ε, να έχουμε μια ε, συνεκτική θέση προς όφελος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ουκρανικού έθνους. Τα κόμματα και οι κυβερνήσεις έρχονται και απέρχονται, όμως οι λαοί παραμένουν ευχαριστώ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ε, θα γίνει η συνάντηση αύριο με τους άλλους ε, σκιώδες εισηγητές και σίγουρα θα γίνει και πάλι εξελόγηση της κατάστασης και νομίζω ότι θα ε, πλησιάσουμε περισσότερο την από Ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης. Ο κύριος Γκάλερ που της αντιπροσωπείας ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Αφρικανική Ένωση θα πάρει το λόγο. Έλαβε χώρα η αποστολή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κύριε Γκάλερ, παρακαλώ, ε, σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, πράγματι. Δεν ακούμε δυστυχώς τον ομιλητή. Πρόεδρε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όντω είχαμε μια αντιπροσωπεία τριών ατόμων στην Αφρικανική Ένωση. Εγώ ήλπιζα ότι θα ήμασταν πιο πολλοί αριθμοί και με καλύπτοντας ένα ευρύτερο πολιτικό φάσμα. Όμως ήταν η πρώτη μας επίσκεψη εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και όχι με τη συνήθη προσέγγιση από την αναπτυξιακή πλέον πρόπτικη. Ε, προσπαθήσαμε να αποτιμήσουμε το ρόλο το όραμα μάλλον της Αφρικανικής ε, Ένωσης ε, για το μέλλον της ως εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θελήσαμε να δούμε τι ανάγκες έχει η Αφρικανική Ένωση στη διαδικασία για την οικοδόμηση δυνατοτήτων και των θεσμικών ε, φορέων. Επίση, τη δυνατότητά τη να προωθήσει την πολιτική ολοκλήρωση και τον εκδημοκρατισμό. Όλα τα στοιχεία αυτά είναι ζωτική σημασία, σημασίας, εφόσον θέλει να είναι ένα σοβαρό εταίρο η Αφρικανική Ένωση, να είναι ένα σοβαρό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναντήσαμε τον Επίτροπο για την Ασφάλεια, κύριο Λαμάμπρα, και τον Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Κουέσα Λάμπα. Και όπω ε, η συνάντηση έγινε στην Αιθιοπία, είδαμε και τον κύριο Μαλισενάου, πρόεδρο τη Αιθιοπική Βουλή, καθώ και πρέσβη τη Αιθιοπία, τη Νότια Αφρική, τη Αλγερία των Αφρικανικών ε, κρατών παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσώπους ε, του ΟΗΕ. Είχαμε μια συζήτηση Τρογγυλή Τραπέζη και με τη συμμετοχή των δικών μα πρέσβεων και του εκπροσωπού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματά μα. Πρώτον, η Αφρικανική Ένωση βραδέω μεταβαίνει από το δυναμικό που διαθέτει προ τα αποτελέσματα, άρα πέραν της οικονομικής στήριξη και των ε, τεχνικών βοηθημάτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία των ε, δυνατοτήτων ε, και την πρόοδο της χώρας, μπορεί επιπλέον να συμβάλλει στην πολιτική σταθεροποίηση και την ειρήνευση στην Ήπειρο με σαφείς όρους. Θα πρέπει να, να συνειδητοποιήσουμε ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τη Αφρικανική Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο να υπάρχει διαρκής συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης ώστε να υπάρχει η ανάληψη ιδιοκτησίας και μάλλον η ανάληψη πρωτοβουλειών και η εντατικοποίηση προσπαθειών. Θα πρέπει η Αφρικανική Ένωση να συνεχίσει τις προσπάθειες χρηματοδότησης και της αυτοχρηματοδότησης. Και εμείς βεβαίω μέσω των κοντελείων του προπολογισμού μας είμαστε ο βασικός χρηματοδότης της Αφρικανικής Ένωσης θεσμικός, ε, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο που πήγαινε από τη Λιβύη, από τον Καντάφη και 17 άλλες χώρες στην Αφρικανική Ένωση, αυτά όλα αλλάζουν αυτά αντικαταστάθηκαν ή πρόκειται να αντικατασταθούν εφόσον η Αφρικανική Ένωση και τα κάτι της μπορέσουν ε, να βελτιώσουν τη συνεισφορά τους. Το καλύτερο θα ήταν να συνεχίσουμε και εμείς το θετικό μας ρόλο. Επίσης, σημαντικό είναι καθώς άλλοι διεθνείς παράγοντες θέλουν να δραματίσουν σημαντικό ρόλο στην Αφρική, εμείς να μην τους ε, παραχωρήσουμε τη θέση μας. Η εταιρική αυτή σχέση και το όραμά μας για την όλη διαδικασία είναι ζωτική συμμαχία. Ενώ η Κίνα πατάει πόδι στην Αφρική όλο και πιο σημαντικά. Υπάρχει ε, η οικοδόμηση της έδρας της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίσα που έχουν αναλάβει κινέζικα κονσόρσια. Για την αφρικανική κρίση επίσης ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ε, μεγαλύτερες προσπάθειες, επικριτικά σχόλια, παρόλο που δεν ήταν από την ε, πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σχόλια, αλλά από τον ΝΑΤΟ που έχουμε και εκεί σοβαρή συμμετοχή, βρήκαμε ότι παραμεριστήκαμε σε σχέση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Αφρική ή προκειμένου να εξυπηρεστούν προβλήματα οι Ευρωπαίοι, μας είπε το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να μην είχατε ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία. Ε, ήμασταν έτοιμοι να διαπραγματευτούμε. Εγώ τους είπα σαφώς και νομίζω αυτή είναι η άποψη και του Κοινοβουλίου μας εδώ ότι είχαμε σαφώς την αίσθηση ότι Εάν στη Βεγγάζη δεν είχε αναλυφθεί άμεσα δράση από τον ΝΑΤΟ όποιους ήταν εκεί, θα είχαν γίνει σφαγές, θα είχαν διπραχθεί σφαγές κατά του πληθυσμού. Τώρα λοιπόν με τη νέα πολιτική κατάσταση στη Λιβύη μπορεί να συνεργαστούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά με την Αφρικανική Ένωση. Ακόμη. Υπάρχει δραστηριοποίηση της Αφρικανικής Ένωσης και προσπαθούν να στο ε, πλαίσιο των διεθνών δυνάμεων στη Σομαλία, της Αμισόμ και της περίπτωσης να επιδεικνύεται πολιτική τους βούληση. Ε, μπορούν να δράσουν φαίνεται εφόσον υπάρχει ανάγκη. Αυτό φάνηκε και σε μια κρίση στην ίδια την Αφρικανική Ήπειρο. Επίσης, αυτό που προέχει είναι οι Αφρικανοί να λύνουν τα προβλήματα της Αφρικής με τον Επίτροπο Λαμάμρα για την Ειρήνη και την Ασφάλεια συζητήσαμε ότι πέραν της οικονομικής και τεχνικής στήριξης για την οικοδόσμηση θεσμικών φορέων και των δυνατοτήτων τους χρειάζονται και περισσότεροι στρατιωτικοί πόροι ώστε η απόκριση της Αφρικανικής Ένωσης να γίνει πιο αποτελεσματική. Ήταν πολύ συγκεκριμένο το θέμα της του προστασίου τους. Τους είχαν, ε, μας είχαν υποσχεθεί πανεπολεμικά ελικόπτερα και επίσης να δημιουργηθεί μια πτήση απαγορεύσης πτήσεων με τη Σομαλία. Στα σύνορα με τη Σομαλία. Αυτό ε, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, τέθηκε ως αίτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θετική απάντηση δεν δόθηκε. Χρειάζονται λοιπόν καλύτερο εξοπλισμό για να μπορέσουν ε, να προστατεύσουν την Υπάρχει λοιπόν περισσότερο περιθώριο για συνένεση μεταξύ των τοπικών ε, οργανισμών στην Αφρική και ανάγκη προσέγγισης όχι μόνο από την κορυφή προς τα κάτω, αλλά και από τα κάτω προς την κορυφή. Αμφίδρομη λοιπόν διαδικασία χρειάζεται για να ενισχυθεί περιφερειακή ολοκλήρωση της Αφρικής. Και οι οργανισμοί που ήδη υπάρχουν έχουν και φιλόδοξη, φιλόδοξο κατάλογο προτεραιοτήτων. Στην επόμενη σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης θα ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία αφρικανική για την δημιουργία ενιαία αγορά. Εν τω μεταξύ, σχέσει συνεργασία με αναβάθμιση των περιφερειακών οργανισμών ενισχύονται διαρκώ και νομίζω ότι θα είναι καθοριστική σημασία για την περαιτέρω ολοκλήρωση. Ο δημοκρατικό έλεγχο παραμένει ένα θέμα. και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και του κοινοβουλευτικού ελέγχου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης καθώς και τη δικασία λήψης αποφάσεων στην ίδια την Αφρικανική Ένωση. Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Είναι γεωγραφικώς εντοπισμένοι, αλλά ε, από πολιτική άποψη ε, στο περιθώριο. Οπότε θα πρέπει να, να τους παρέσχουμε ακόμη περισσότερη πολιτική, περισσότερη πολιτική στήριξη. Για να ενισχυθεί ο ρόλος του στην Αφρικανική Ένωση. Δημερός στην Αιθιοπία συναντήσαμε τον Πρωθυπουργό και για να το πω απλά είναι σκληρός τύπος. Είναι πραγματικά σκληρό καρύδι. Ε, και με μια κυβέρνηση στο ευάλωτο κέρας της Αφρικής πραγματικά διδραματίζουν ρόλο σταθεροποιητικό σε σχέση με άλλους ε, γειτονές τους στην περιοχή. Πραγματικά η Αιθιοπία εξισορροπεί την κατάσταση. Και παρόλα αυτά δεν είμαστε καπνοποιημένοι με τη δημοκρατική τους αγωγή. Να θυμίσω ότι για δεύτερη φορά μετά το 2005, το 2010, είχαμε ε, αποστολή παρατήρησης εκλογών Όμως δεν μπόρεσε ο εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει την τελική του έκθεση. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν είπε ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, θα πρέπει λοιπόν να καταγράψουμε τις συνέπειες. Και έδωσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με ένα μνημόνιο συνεννόησης, όπως αυτό που είχαμε ετοιμάσει για την Τινησία με την τότε αποστολή μας παρατήρησης. Ε, είχαμε ζητήσει από τον επικεφαλής παρατηρητή να παρουσιάσει την τελική έκθεση κατά την επιστροφή μας. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Αιθιοπία. Για να ολοκληρώσω. Ο ρόλος μας ως Ευρωκοινοβουλίου. Νομίζω θα πρέπει να αναζητήσουμε στήριξη να παράσχουμε μάλλον θεσμική στήριξη στην Αφρικανική Ένωση ως ε, στοιχείο διευκόλυνσης για την οικοδόμηση δυνατοτήτων και θεσμικών φορέων. Βάσει αυτή τη στήριξη θα πρέπει να είναι όροι και προποθέσει, ε, επιδόσει και λογοδοσία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο βασικό δωρητή. Επίση, θα πρέπει επιπλέον, ε, καθότι αυτό είναι αποτελεσματικό σε κάποιες περιοχές, πέραν της τεχνικής ε, υποστήριξης περιφερειακών οργανισμών ε, στην Αφρικανική Ένωση, να πράγουμε και το ρόλο τους για την, δημοκρατικό και περιφερειακό, για την δημοκρατική και περιφερειακή ολοκλήρωση. Πολλοί από τους συνομιλητές μας ζήτησαν ε, μια παναφρικανική οικονομική ένωση ώστε να ασχοληθεί με τις οικονομικές ανάγκες της Αφρικανικής Υπήρου. Το συζητήσαμε και στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης το Δεκέμβριο και οι συνάδελφοί μας από την Αφρικανική πλευρά είπαν υπάρχει ανάγκη να ξεπεράσουμε την φιλοσοφία της ΑΚΕ. Ξέρουμε τις συμφωνίες της Κοτονού και τις μορφές συνεργασίας που καθορίζουν Σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίζει ως ενίο σύνολο την Αφρική. Αυτός ό,τι αφορά την πολιτική τη προσέγγιση. Η διπλή ταχύτητα λοιπόν από τη μια η κοτονού από την άλλη αφρικανική στρατηγή θα πρέπει να συζητηθούν ώστε να μπουν στην ίδια την ε, πορεία. Τέλος, δημοκρατικός διάλογος με την Αφρικανική Ένωση για τις πολιτικές της επιλογές και με προπρόθεσμα δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης και σύστημα δημοκρατικού διαλόγου και δημοκρατικού, δημοκρατικής λογοδοσίας. Εύχομαι εμείς ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να διατηρήσουμε σε αιτήσια βάση τις επαφές μας με την Αφρικανική Ένωση για τον επιπλέον λόγο ότι έχουμε να κάνουμε με μια ήπειρο σε κρίση. Κάποιοι είναι και γειτονέ μας. Δεν αφορά λοιπόν αυτό μόνο την εξωτερική μας πολιτική. Κάποιοι άλλοι λίγο μακρύτερα επηρεάζουν τους κοντινούς. Και εμάς εδώ. Πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε τα θέματα αυτά και ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε. Well, thank you. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε εικόνα το πώς, βλέπουν, πώς βλέπει τα πράγματα η άλλη πλευρά. Η πρόταση αυτή να προσπαθήσουμε να αποκατηστήσουμε μια ετήσια επαφή μαζί τους είναι καλή. Επιθυμεί κανείς να προσθέσει ή να ρωτήσει. Αν όχι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλερ. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο μεταξύ 12 και 30 και 13 και 45 θα είναι μαζί μας ο κύριος Φίλε